Συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ελπίζω να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο με την αργία, όσοι δεν είχαν την αργία. Είναι φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία λοιπόν, εγκρίνεται. Στις ανακοινώσεις του Προέδρου τώρα. Να σας υπενθυμίσω και πάλι διάφορες εκδηλώσεις της Επιτροπής μας. Καταρχάς ένα εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Αντίδραση στις ε, καταστροφές αύριο το απόγευμα, European Disaster Response, είμαστε αρμόδιες και σε τέτοιες, για τέτοιες περιπτώσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να είναι έντονο το ενδιαφέρον και η συμμετοχή μας στο εργαστήριο αυτό. Στις 21 Ιουνίου έχουμε μια ακρόαση για τη Βαλτική. Στο, στο, στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής μας και σε αυτό σας συστήνω να συμμετάσχετε και ένα εργαστήρι για την αλλαγή του κλίματος και για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις 8 Ιουνίου από τις 4 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Για την προστασία του κλίματος, σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στην Βόνη, δεν έχω κάτι να σας αναφέρω. Όπως πάντα στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ όποια πρόοδος ε, σημειώνεται, σημειώνεται στην τελευταία στιγμή. Προς το παρόν έχουμε μάλλον τελμάτωση και δυστυχώς όχι μεγάλη πρόοδο, αλλά ακούσαμε από την Διεθνή ε, Υπηρεσία Ενέργειας πώς αυξήθηκαν τα ποσοστά εκπομπών τα τελευταία έτος 30,6 γιγατόνους. Σκοπός μας ήταν να είναι πολύ πιο χαμηλό αυτό το ποσό. Άρα έχουμε σημειώσει καθυστέρηση. Να σας ανακοινώσω κάτι καινούριο, μία είδηση. Ο συνάδελφος Κυλακάκης άλλαξε πολιτική ομάδα. άφησε την ε, μεγάλη ομάδα και μεταπίδησε στην ομάδα Άλτε, στους φιλελεύθερους, ο συνάδελφος Κυλακάκης. Ανήκει πλέον στην ομάδα των φιλελευθέρων. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά θα ερευνήσουμε κατά πόσον μπορεί να σημαίνει κάτι για τους βαθμούς εδώ στην Επιτροπή μας. Ωραία. Και περνάμε στο πρώτο σημείο επί της ουσίας, στο 3. Έλεγχος των κινδύνων που συνδέονται με τα μείζωνα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες. Γιάννος Άντερ, ο συζητητής, ο οποίος έχει ερευνήσει το, το θέμα αυτό, αλλά να προτείνω να καλέσουμε καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την οδηγία αυτή, την οποία δεν έχει παρουσιάσει ακόμα εδώ. Εργάζεται ωστόσο στο θέμα αυτό ήδη η κυρία Μαριάννα Βένινγκ από την Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ. Αν θα θέλετε λοιπόν να πάρετε το λόγο για να μας εξηγήσετε τι, ποιος είναι ο σκοπός της ε, οδηγίας. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Ως, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα σας παρουσιάσω εν συντομία το έργο μας. Να πω ότι είμαστε ευγνώμονες προς την Επιτροπή και ιδιαίτερα προς τον κύριο Άντρη για την δουλειά που έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε να δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα ε, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα σχολιάσω ακόμα την, ε, το έργο του κυρίου Άντερ. Θα περιοριστώ στην σύντομη παρουσίαση της οδηγίας. Να σας υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε η διαδικασία το 2008 λόγω της ανάγκης να αναρμονιστεί ο ορισμός ε, ε, των επικίνδυνων ουσιών με τις ισχύουσες προσδιαγραφές. Αυτά που αναφέρονται στην ε, λεγόμενο κανονισμό ACP που ρυθμίζει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εναρμονισμένο σύστημα για την κατάταξη των χημικών ουσιών. Οι βασικές διατάξεις της οδηγίας ουσιαστικά παραμένουν απαραλλακτές από το 1996 που εγκρίθηκε. να αναθεώρηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσο ε, θα έπρεπε να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις στην οδηγία. Τα καλά νέα είναι ότι η τρέχουσα οδηγία περιόρισε πάρα πολύ τα ατυχήματα και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους. Ωστόσο, στην τελευταία εκτίμηση της οδηγίας και των περιστατικών βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε 20 με 35 μεγάλα ατυχήματα τα οποία αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει φυσικά να γνωρίσουμε ότι αυτό είναι μεγάλος αριθμός ατυχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν σκοπός μας να είναι η περαιτέρω μείωση αυτών των μεγάλων ατυχημάτων και των συνεπειών τους και να προσαρμοστεί φυσικά ανάλογα και το αριθμιστικό πλαίσιο. Προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια απλή λύση για να εναρμονιστούμε απόλυτα με το νέο σύστημα εναρμόνισης ε, κατάταξης που αποτελεί άλλωστε και το βασικό σκόπο του εγχειρήματος. Σκοπός μας είναι να διατηρηθεί το επίπεδο προστασίας και εκ να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στο εύρος εφαρμογής της οδηγίας. Θεωρούμε ότι έχουμε βρει μια σωστή ισορροπία. Επειδή οι μελλοντικέ αλλαγές ε, για την κατάταξη των χημικών ουσιών θα ε, επηρεάσει την εφαρμογή της οδηγίας, έχουμε συμπεριλάβει και έναν μηχανισμό διόρθωσης για να περιορίσουμε ανεπιθύμητες ε, παρενέργειες, αν θέλετε, αυτών των αλλαγών. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται στο έυρος, στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία σε βέζο κάποιε ουσίε ανάλογα με τον ενδεχόμενο κίνδυνο που ε, παρουσιάζουν. Για να βελτιωθεί ε, επίσης και το επίπεδο προστασίας. Θεωρούμε ιδιαίτερα ότι η η δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και η επιθεωρήση αποτελούν βασικές διατάξεις προς αυτή την κατεύθυνση και αυτές οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να βελτιωθούν. Προτείναμε βασικές πληροφορίες για τον κίνδυνο και για την ασφάλεια και η σωστή αντιμετώπιση ενδεχόμενου ατυχήματος θα πρέπει διαρκώς μέσω διαδικτύου να παρέχονται στο κοινό. Και θεωρούμε ότι είναι σωστή αυτή η πρόταση. Επίσης, οι πιο λεπτομερείς κανόνες και οι συγκεκριμένες διατάξεις για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους. Και θεωρούμε λοιπόν ότι η οδηγία συνάδει πιο πολύ με τις στόχους του άρχους. Επίσης, ε, προτείνουμε πρότυπα για την επιθεώρηση και τον έλεγχο συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων συχνότητας που των ελέγχουν αυτών. Πρόεδρε, ελπίζω να είναι επικοδομητική η συζήτησή μας και να είναι και στενή συνεργασία μας με την Επιτροπή σα και με το Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βένινγκ, για την παρουσίαση αυτή της οδηγίας σε Βέζο 3. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Άντερ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Η κυρία Δένιγκ ε, με διευκόλυνε, διότι παρουσίασε πάρα πολύ ξεκάθαρα το στόχο αυτής της πρότασης. Μας ανέφερε πολύ καλά το τι έγινε τους τελευταίους μήνες και γιατί παρουσιάστηκε η πρόταση για τροποποίηση της ΕΒΕΖΟ 2. Η κυρία Δένινγκ επίσης ανέφερε ότι στο παρελθόν έχουν εγκριθεί σχετικές διατάξεις σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εναρμονίσουμε αυτές τις δύο διατάξεις. Και αυτό είναι και ο λόγος που μας οδηγεί να σας αναφέρω εδώ ότι γιατί τροποποιούμε την οδηγία έπαιζο. Στόχος μου ήταν να μπορέσω να διασφαλίσω τη συνοχή των διατάξεων. Δεύτερος στόχος μου ήταν πολιτικός, να διατηρήσουμε δηλαδή τουλάχιστον το τωρινό επίπεδο ασφάλειας. Και τρίτος στόχος, τα ήδη λιμένα προβλήματα σε επίπεδο παλαιών διατάξεων δεν πρέπει να ξανασυζητηθούν. Αυτό ισχύει και για τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία επίσης δεν τα αμφισβητούμε. Επίσης, θα ήθελα να σας αναφέρω πώς συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους τους τελευταίους μήνες συναντήσαμε εκπροσώπους ε, από την Κομισιόν, από τη βιομηχανία, από τα, από τα λόμπις κλπ. Έγινε μια ακρόαση τελικά με εκπροσώπους του Συμβουλίου, της Κομισιόν, των εκπροσώπων του κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών και όλοι μπόρεσαν να εκφραστούν για το θέμα η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, μιλάω για αυτήν της 13 ε, Απριλίου. Απριλίου, είχαμε μετά συναντήσεις με τους σκεώδεις εισηγητές. Και μαζί αναζητήσαμε τα πιο σημαντικά σημεία της όλης προβληματικής όπως επίσης αναζητήσαμε και συμβιβαστικές λύσεις για να γεφυρώσουμε εκεί όπου είχαμε τις μεγαλύτερες διαφορές. Οι τροπολογίες που κατέθεσα είναι καθαρά ε, μερικές τεχνικού χαρακτήρα και άλλες καθαρά περιεχομένου. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στις τροπολογίες τεχνικού χαρακτήρα, αλλά να σταθώ στις τροπολογίες ουσίας. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου να αναφέρω στην Κομισιόν και στους συναδέλφους ένα σημείο. Για το παράρτημα 1 εγώ δεν έχω παρουσιάσει καμία αλλαγή γιατί είχαμε, έστω και αν είχαμε πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό. Εγώ υποστηρίζω τη θέση της Κομισιόν. Οι εκπρόσωποι όμως της βιομηχανίας και άλλων πολιτικών ομάδων παρουσίασαν εντελώς διαφορετικές θέσεις. Μετά από την τροποποίηση της οδηγίας ΕΒΕΖΟ 2, αναρωτιέται κανείς Ποιος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται, καλύπτονται από το εφαρμοστικό πεδίο της οδηγίας έμπεζου. Είναι γύρω στις 10.000 επιχειρήσεις. Η κατάσταση όμως είναι εντελώς ετερογενής. Εμείς ακούσαμε διάφορες εκτιμήσεις από τη βιομηχανία που λένε ότι σήμερα αυξάνονται κατά 30% οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες ε, οι οποίες εντάσσονται στο εφαρμοστικό πεδίο. Η Κομισιόν όμως λέει όχι, ίσα ίσα μειώνεται κατά 2% το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων. Και μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Ο αριθμός των επιχειρήσεων επικινδύνων ουσιών ε, έχει αυξηθεί. Άρα έχουν αυξηθεί κατά συνέπεια και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Άρα εμείς πρέπει να δεχθούμε μία αύξηση του 3% που και η κυρία Βένιγκ λέει 3% είναι κάτι το αποδεκτό. Εμείς όμως συνεχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε σε τι οφείλεται αυτό, αυτή η τεράστια διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ της βιομηχανίας και της Κομισιόν. Ίσως το γεγονός ότι η βιομηχανία δεν λαμβάνει υπόψη της ότι πολλές από αυτές τις επικίνδυνες ουσίες ε, αφορούν σε πυροελάχιστες ποσότητες στα εργαστήρια ορισμένων εργοστασίων, οπότε δεν εμπίπτουν μέσα στο εφαρμοστικό πλαίσιο της οδηγίας. Κάτι άλλο το οποίο δεν θεωρήθηκε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέες ουσίες οι οποίες καταλήγουν στον κατάλογο παράγονται από επιχειρήσεις οι οποίες ούτως ή άλλως εντάσσονταν στο εφαρμοστικό πεδίο της ΕΒΕΖΟ 2. Και ίσως σήμερα απλώ παράγουν μια-δυο ουσίες παραπάνω. Δηλαδή είπαμε επιχειρήσεις που με το παλιό καθεστώς επίσης καλύπτονταν. Κοιτάω την ώρα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Αν έχετε αναλυτικές ερωτήσεις τότε και εγώ να σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως. Για τις τροπολογίες θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν, το θέμα των παρεκκλήσεων και των εξουσιοδοτημένων πράξεων. Εγώ έχω μία διαφορετική άποψη από αυτή της Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι όλοι σας έχετε μία... Έχετε αναλυτικά το, το, έχετε το κείμενο μπροστά σας, τουλάχιστον στα αγγλικά. Εγώ πιστεύω ότι η τροποποίηση του παραρτήματος 1 μπορεί να προκύψει μόνο μέσα σε πλαίσιο συναπόφασης. Θα πρέπει όμως να αφήσουμε και στην Κομισιόν τη δυνατότητα να εφαρμόσει ορισμένες δυνατότητες παρεκκλήσεων, όπως επίσης και τα κράτη-μέλη, αν φυσικά το θεωρούν σωστό ότι μία συγκεκριμένη οδηγία θέλουν να μπει στον κατάλογο της οδηγίας σε βέζο, να μπορούν να το κάνουν. Εγώ κατέθεσα τις τροπολογίες μετά από συναντήσεις με τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών ομάδων και υπάρχει και ένα άλλο αντιμαχόμενο σημείο που αφορά στην κοινή γνώμη. Εγώ έχω μία διαφορετική θέση από αυτήν της Κομισιόν. Θα παρακαλούσα στους συναδέλφους να κοιτάξουν να προσπαθήσουν μάλλον να κατανοήσουν τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή μου τη θέση. Εισαγωγικά θέλω να πω ότι Φυσικά και συμφωνώ απόλυτα με το στόχο ουσίας ε, της Κομισιόν. Όσον αφορά όμως στην εμπλοκή των περίοικων σε όλη αυτή την ιστορία θεωρώ ότι οι περίοικοι των εργοστασίων θα πρέπει να έχουν απόλυτη διαφάνεια, θα πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα και σε περίπτωση δυστυχήματος θα πρέπει να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και μέσω ίντερνετ πρέπει να δίνονται αυτές οι πληροφορίες. Θα ζητούσα επίσης από τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη τους ένα άλλο ζήτημα. Ε, εντάξει οι πληροφορίες να δίνονται στο διαδίκτυο φυσικά Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι, κίνδυνοι και σε θέματα ασφάλειας. Με επιπτώσεις στην ίδια την παραγωγή των εργοστασίων αυτών. Ορισμένες τεχνικές πληροφορίες θα μπορούσαν ίσως να μπερδέψουν περισσότερο από ότι να πλουστεύσουν την πληροφόρηση η παραγωγή χημικών ουσιών που, μπορεί, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μπορεί να ε, αποτελούν κίνητρο και για τρομοκράτες. Ε, πρέπει αυτά να βρίσκονται στο ίντερνετ και αυτές οι πληροφορίες να είναι ανοιχτές σε όλους και όχι μόνο στους περίκους. Μετά έχουμε τους ελέγχους, τους επιτόπου ελέγχους. Κατά τη γνώμη μας, πάνω από τις μισές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Σέβεζο 2, εμπίπτουν και στην οδηγία εκπομπών επικινδύνων ουσιών. Θα έλεγα λοιπόν να ενοποιήσουμε τους ελέγχους ακριβώς για να απεισχνεύσουμε την όλη διαδικασία. Συγγνώμη πρόεδρε που μακρηγορώ, αλλά ε, και που εκμεταλλεύτηκα το χρόνο σας, αλλά δεν τα πακαν όλα. Οπότε αν χρειάζονται διευκρινήσεις θα απαντήσω πάρα πολύ ευχαρίστως. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ αντικαθιστώ τον Τζον Λάινεν που θα επανέλθει αργότερα γιατί είχε κάποια συνέντευξη να δώσει. Και τώρα θα ακούσουμε του σκιώδεις εισηγητέ. Να σα ευχαριστήσω εσά για την εισηγησή σα. Πρώτο. πρώτη, η κυρία Βέσλοντ, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Άντερ για τις πολύ επικοδομητικές συσκέψεις που είχαμε μέχρι στιγμής ε, με πολύ ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας. Έχουμε συναντηθεί μέχρι στιγμή Να καλωσορίσω την έκθεσή σα. Σα υποστηρίζω στα όσα προτείνεται για εναρμονισμένα κριτήρια για εξαιρέσει ε, και ότι αυτά θα επιφασιστούν μέσω νομοθετική πράξη. Πιστεύω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό κέριο κομμάτι αυτής της νομοθεσίας και θα πρέπει να περάσει από συναπόφαση. Επίσης συμφωνώ με τον κύριο Άντερ και όπου λέει ότι οι εξαιρέσεις που χορηγούνται από τα κράτη-μέλη με ορισμένου όρου, θα πρέπει να αφορούν μόνο τις συγκεκριμένε διατάξεις και ότι η θέσπιση τους ε, θα αφορά την ε, θέσπιση ε, ε, κατώτατων όριων. Νομίζω πως με αυτό συμφωνούμε και στο Κοινοβούλιο και με βάση τα όσα έχει πει μέχρι στιγμής η Κομισιόν. Ωστόσο, δεν υποστηρίζω τις αλλαγές του κ. Άντερ στην πρόταση της, κυρίας, της Κομισιόν όσον αφορά την ενημέρωση. Πιστεύω πως η Κομισιόν έχει κρατήσει ισορροπημένη στάση και γραμμή και δεν πιστεύω πως μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στην ενημέρωση που έχουμε από το ίντερνετ και τα όσα μπορεί κανείς να έχει ως πολίτης, υποστηρίζοντας ότι οι τρομοκράτες μπορεί εύκολα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στο ίντερνετ. Ο τρομοκράτης ούτως ή άλλως μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Άρα λοιπόν πιστεύω πως θα πρέπει να διατίθενται στο ίντερνετ οι πληροφορίες αυτές γιατί ε, μόνο έτσι μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Υποστηρίζω λοιπόν τη θέση της Κομισιόν από αυτού. Έχω κάποιες τώρα αμφιβολίες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Ε, νομίζω πως θα προτιμούσα να συμπεριληφθούν οι αγωγοί εδώ καθώς και οι πλατφόρμες εξόρυξης. Νομίζω πως, ξέρω μάλλον πως προετοιμάζονται σχετικές νομοθεσίες, νομοθετικές προτάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν τις έχω δει. Γι' αυτό και κάπου θα πρέπει να περιληφθούν και όλα αυτά. Και αυτή είναι η νομοθεσία, που, η νομοθετική πρόταση που εξετάζουμε τώρα. Για την άμεση αποθήκευση, πράγμα το οποίο συζητήσαμε και στις συσκέψεις μεταξύ σκιωδών συγητών, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογή μέχρι στιγμή. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο καιρό μπορεί κανείς να αποθηκεύσει κάτι πριν πριν να χρειαστεί ή μάλλον πριν να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής. Αυτή είναι ερώτηση προς την Κομισιόν μάλιστα. Πόσο καιρό μπορεί κανείς να αποθηκεύσει κάτι πριν να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής. Επίσης, όταν ευθυγραμμίζεται το παράρτημα 1 στο κανονισμό CLP, το αποτέλεσμα κάποιες φορές είναι αμφισβητήσιμο. Για παράδειγμα, φαίνεται να χαμηλώνει το επίπεδο προστασίας για τις διοξίνες, προστασία για τον άνθρωπο αλλά και για το περιβάλλον, ε, θα ήθελα λοιπόν αυτό να το, να το εξετάσω περισσότερο πριν αποφασίσω και τέλος θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Κομισιόν γιατί αποκλεί την ε, ε, στοματική έκθεση. Έχουμε στοιχεία για αυτά όλα και η έκθεση ε, η στοματική μέσω της κατάποσης νερού ε, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θα πρέπει να μείνει εκτός λοιπόν. Αυτή είναι ερώτηση, ακόμα μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον Παναγιώτοφ από τους φιλελεύθερους εδώ. Μπορείς θέλει κάποιος άλλος από τους φιλελεύθερους να πάρει το λόγο. Όχι τότε θα μου δώσω το λόγο εγώ γιατί είμαι σκιώδης για τους πράσινους. Ε, σας ευχαριστώ για τη σπουδαία σας εργασία. Είχαμε πράγματι πολύ πικοδομητικές ε, συναντήσεις. Καλωσορίζω και συμφωνώ με την έκθεσή σας. Ε, έχω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις και εγώ ανησυχώ όσον αφορά τις τροπολογίες για τη διαφάνεια Έχουμε 30 μεγάλα ατυχήματα ετησίω με τέτοιου είδου εγκαταστάσει και μέχρι στιγμής δεν είχαμε ούτε μια τρομοκρατική επίθεση κατά τέτοιου είδους ε, εργοστασίων. Νομίζω ποτέ μάλιστα δεν έχει γίνει τρομοκρατική επίθεση, οπότε ε, από ό,τι βλέπουμε και από την ε, μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν, βλέπουμε πως ε, το, η διαφάνεια είναι το ασφαλέστερο μέσο ασφάλειας που μπορούμε να έχουμε. Νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι ωφέλιμο τόσο από άποψη οικονομική όσο και για λόγους ασφάλειας. Έπειτα, δεν χρειάζεται να είναι κανείς χημικός μηχανικός για να γνωρίζει ποιες ουσίες ε, χρησιμοποιούνται σε ποια εργοστάσια ούτως ή άλλως. Άλλα θέματα τώρα. Κάπως με ανησυχεί η λογική που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για την μη αύξηση του αριθμού των ε, εγκαταστάσεων και των εργοστασίων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσες, πόσες εργοστάσια καλύπτονται. Το σημαντικό είναι να καλύπτονται ε, τα επικίνδυνα εργοστάσια. αυτό είναι το ζήτημα, γι' αυτό κάνουμε αυτή την νομοθεσία. Αν είναι 5% παραπάνω ή 2% λιγότερες, δεν μας ενδιαφέρει. Το σημαντικό είναι η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της οδηγίας. Δεν πρέπει να φέρουμε λοιπόν κατηγορίες από αυτόν τον κατάλογο μόνο και μόνο για να έχουμε τον ίδιο αριθμό εγκαταστάσεων εργοστασίων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και έπειτα το, ποιες αριθμός μάλλον των εγκαταστάσεων που καλύπτονται θα εξαρτάται από τι είδους παραγωγή εκάνουν έχουν. Επίσης, για την ενδιάμεση υποθήκευση είναι σημαντική και οι εξαιρέσει από την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μια επικίνδυνη ουσία που προετοιμάζεται ε, είναι επικίνδυνη μονίμως. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε συνολική δηλαδή εξαίρεση για τις πλατφόρμες εξόριξης ανοιχτής θαλάσσης. Αυτές οι εξαιρέσεις λοιπόν θα πρέπει να αφαιρεθούν, θα πρέπει να εξεταστούν όπως και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις, εργοστάσεις. Αν υπάρχει κίνδυνος ή πιθανός κίνδυνος θα πρέπει να εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας για την κοινοποίηση, άρθρο 6, ε, g και άρθρο 8. Είναι δύσκολο αν ένας ε, φορέας ευέζο δεν έχει πληροφορίες για τις ε, ουσίες που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη δική του την ίδια την ασφάλεια είναι δύσκολο. Ίσως θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να κάνουν αξιολογήσεις και για τις γειτονικές, τα γειτονικά εργοστάσια για να μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες και για το άρθρο 19 νομίζω πως είναι πιο λογικό να έχουμε ετήσια επιθεώρηση και για τα εργοστάσια του χαμηλότερου στρώματος γιατί διαφορετικά ε, θα αντιμετωπίζονται όπως σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία σε φέζο. Τώρα, το όριο του ενός κιλού δεν είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Καλύτερα είναι να έχουμε ένα κατόφλι συνδυασμού μεταξύ βάρους και ε, πυκνότητας. Μέχρι στιγμής έχουμε δουλέψει πολύ καλά για αυτό το θέμα ε, και γι' αυτό και περιμένω και την ε, συνεργασία μας και για την ολοκλήρωση. επόμενη ομιλή, ομιλήτρια είναι η Σαμπίνε Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για τη συνεργασία και για το κλίμα το οποίο επικράτησε στις συναντήσεις με τους κοιόντες συζητητές. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην μειωθεί το εφαρμοστικό πεδίο. Με τη ΣΕΒΕΖΟ 3 θα πρέπει να ενισχύσουμε τον παράγοντα ασφάλεια και να τον επεκτείνουμε. Πρέπει να εγγυάται η οδηγία την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους πολίτες και για την κοινωνία. Οι καρκινογόνες χημικές ουσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο 1. Όπως επίσης και οι ουσίες εκείνες οι οποίες δημιουργούν μακροχρόνιες βλάβες και τα CCS. Πρέπει επίσης ε, να καταγραφούν διότι πρόκειται για τεχνολογία η οποία ενηχεύει κινδύνους. Δεν έχουμε παρκής γνώσεις για το θέμα των offshore για τις πλατφόρμες ε, ε, offshore για τους σταθμούς, θυμηθείτε τι έγινε με το συνδρομικό δυστύχημα στο Βιαρέτζο. Με τις χωματερές, όλα αυτά θα πρέπει να τα καλύψουμε. Θα πρέπει η τροποποίηση του παραρτήματος 1 να περνάει με την συναπόφαση. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τον εισηγητή. Τώρα, για το κατά πόσο θα πρέπει να είναι ανακατεμένη η κοινή γνώμη. Στην όλη διαδικασία της πληροφόρησης. Η Κομισιόν ε, σε αυτό θέτει περιορισμούς ε, στην πληροφόρηση για θέματα ασφάλειας ή για θέματα μυστικότητας, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να επικαλεστεί λόγους για να μην δώσει πληροφορίες. Η κοινή γνώμη θα πρέπει να έχει πληροφόρηση σαφέστατη για τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες αποθηκεύονται κοντά στα σπίτια τους. Το ίδιο και για τα μέτρα ασφάλειας και για τους κινδύνους. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Ούτε καν και οι συνδέσεις με άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή. Εβδομάδες μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα διαπιστώνουμε το πώς ο διαχειριστής του εργοστασίου είπε ψέματα και στην κυβέρνηση και στο λαό για το μέγεθος της καταστροφής. Εντάξει, πρόκειται για ακραία περίπτωση. Αλλά όλες οι πληροφορίες μετά από καταστροφή πρέπει να ανακοινώνονται στην κοινή γνώμη. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέγεται ότι είναι πολύ πολύπλοκες όλες αυτές οι πληροφορίες για να γίνουν κατανοητές από την κοινή γνώμη. Ε, μα αυτό δεν είναι σοβαρό. Τι επιχείρημα είναι αυτό, δηλαδή ποιος έχει το δικαίωμα να κρίνει κατά πόσο ο λαός είναι φύση ή όχι. Και ποιο είναι το επίπεδο ευφύα. Άμα δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση δεν θα έχουμε και σωστή αποτελεσματικότητα της ΕΒΕΖΟ 3. Αυτά δεν πρέπει λοιπόν να υπόκεινται σε εμπορικά κριτήρια. Σύμφωνο με την Κομισιόν για τη βούλησή της να βελτιώσει την οδηγία. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Χρειάζονται όμως και επιπλέον έλεγχοι. Έλεγχοι απρόβλεπτοι. Επόμενο χιλιάδος είναι ο κύριος Ρώση, αλλά δεν τον βλέπω. Ντερώσε, συγγνώμη, αλλά δεν τον βλέπω. Ο πρώτος στον κατάλογο των ομιλητών τώρα είναι ο Καλ Χάινς Φλόρεντς. Ε, kann eigentlich nur sein, dass die Dame der Kommission, als auch unser Kollege Ader, ja so. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν και ο εισηγητής μας έδωσαν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες και κάλυψαν την ουσία Γι' αυτό δεν έχω πολλά να πω. Αλλά παίρνω βέβαια τις αποστάσεις μου από την προλαλή σας συνάδελφο η οποία θέλει να πετάξει το μωρό μαζί με το νερό του μπάνιου. Θέλω να ρωτήσω όμως την Κομισιόν τι κάνουν τα κράτη-μέλη με την υπάρχουσα οδηγία σε Εγώ απαγοητεύομαι τα μάλα κάθε φορά που συζητάμε εδώ για αλλαγές διατάξεων διότι πριν αρχίσουμε να μεταρρυθμίζουμε τις υπάρχουσες διατάξεις πρέπει να δούμε τα κράτη-μέλη τι κάνουν ήδη με την εφαρμογή των υπαρχόντων κανονισμών. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση σε αυτό. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ. Α, υπάρχει αντίχηση. Σε τι να οφείλεται άραγε, λέει ο κύριος Κράμερ, Μπορεί να είμαι ίσως ραδιενεργός, λέει ο κύριος Κράμερ. Αντίστοιχη ερώτηση με αυτή του Φλόρεντς. Προστασία των πολιτών. Σύμφωνοι. Η προστασία όμως δεν θα πρέπει να χειραγωγείται. διότι η προστασία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να επεκτείνουμε το εφαρμοστικό πεδίο σε όλες τις τοξικές ουσίες. Διότι αυτό σημαίνει ότι, όπως είπε και ο Καρχάιντς Φλόρεντς, πετάμε το μωρό μαζί με το νερό του μπάνιου. Ρωτώ την Κομισιόν. Έχουμε μία αποτελεσματική οδηγία σε έπαιζο. Έχουμε γύρω στις τα 30 καταγεγραμμένα δυστυχήματα Και αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα για να προσαρμόσουμε το εφαρμοστικό πεδίο. Ρωτώ όμως, σε τι οφείλονται αυτά τα αντιστοιχήματα, επρόκειτο για εργοστάσια τα οποία δεν καλύπτονται από την Σεβέζο 2 ή καλυπτόντουσαν αυτά τα εργοστάσια. Οι ουσίες ήταν ουσίες που υπάρχουν στην τωρινή οδηγία ή όχι. Αναρωτιέμαι αν η επέκταση του εφαρμοστικού πεδίου κυρίως για την κατηγορία κινδύνου 3 θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε πλεονεκτήματα από πλευράς ασφάλειας. Δεν έχει απαντηθεί το ερώτημά μου ακόμα. Η απορία μου παραμένει μήπως πρόκειται απλώς για γραφειοκρατική φόρτωση των δαπανών. Αν μιλάμε εμεί για 5% ή 30% παραπάνω εργοστασίων που πρέπει να καλυφθούν, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια που δεν έχουμε μεγάλες χημικές βιομηχανίες, παρόλα αυτά, με μία τέτοια οδηγία θα αυξηθούν οι επιχειρήσεις αυτές. Ποια θα είναι η σχέση μεταξύ κόστους ωφέλειας ή θα έχουμε μόνο εμείς μία φόρτωση του γραφειοκρατικού πεδίου. Εκπλήσωμε λοιπόν. Πού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτηνε τον τομέα εφαρμογή για τις συναντήσεις πριν, την από, πριν από την ομάδα δεν είχε διαφανεί καμία τέτοια ένδειξη και έχω το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη να επεκταθεί το τομέα εφαρμογή. Αυτό ω βασικό στοιχείο. Θα ήθελα να αναφέρω ακόμα δυο άλλα ζητήματα στα οποία δεν θα επιμείνω. Η εμπειρία μα ε, από άλλε νομοθεσίε μα καταδεικνύει ότι ο αριθμό των ελέγχων και των επιθεωρήσεων δεν είναι απαραίτητα συνδεμένο με την ασφάλεια. Όχι, αυτό ο αριθμός των επιθεωρήσεων έχει να κάνει με τον κίνδυνο που ενέχει κάθε εγκατάσταση. Οι συχνοί έλεγχοι δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον βαθμό ασφάλειας της κάθε εγκατάστασης. Το θέμα είναι και οι πόροι, το προσωπικό, γιατί είναι εύκολο να προδιαγράφεται η αύξηση του αριθμού, του αριθμού ελέγχων, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο αυτό μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, διαφάνεια, φυσικά και χρειάζεται διαφάνεια, αλλά η δημοσίευση στοιχείων θα πρέπει να ρωτηθούμε μας αποδίδει τελικά ασφάλεια ή μήπως δημιουργεί μια γενικότερη ανασφάλεια αν δεν προσέξουμε γιατί σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τη μεταφορά, η αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Αυτό ε, είπαν κάποιοι ότι μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένες επιθέσεις. Το ότι δεν έχει γίνει αυτό ακόμα είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να προσέξουμε γιατί οι πληροφορίες αυτές ε, όντως ε, που θα δημοσιεύουμε σκοπό θα έχουν τη δημιουργία διαφάνειας ή μήπως θα δημιουργούν επιπλέον κινδύνους με άτομα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις πληροφορίες και ίσως να είναι αντιπαραγωγική τελικά η δημοσίευση. Αυτά ήθελα μόνο να αναφέρω ως σημεία κριτική σε αυτά τα τρία στοιχεία. Κατά τα άλλα να συγχαρώ τον εισηγητή. Τουλάχιστον η έκθεση πραγματεύεται την ουσία του θέματος. Thank you. And, uh... Σας ευχαριστώ. Βλέπω πως είναι εδώ η κυρία Κάτελεν Γκαράν Νάγκη από το Συμβούλιο. Θα θέλατε να πείτε κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Βρίσκομαι εδώ αντιπροσωπεύοντας την Ουγγρική Προεδρία. Προείδρευσα των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας, εάν θέλετε αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να, συγχαρώ τον κύριο Άτερ για την ε, περιστατωμένη του έκθεση και ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε με την Επιτροπή σας και με το Κοινοβούλιο και καρποφόρες διαπραγματεύσεις, αν όλα πάνε καλά. Ε, να σας πω ότι... Ξέρετε πως αυτή η πρόταση δημοσιεύθηκε και εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Ήταν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Η Προεδρία μας θεώρησε πως είναι πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό και το εξετάζουμε από την αρχή της Προεδρίας μας. Το έχουμε ήδη εξετάσει πέντε φορές στην ομάδα εργασία στην πρωτοναρχική πρόταση της Κομισιόν και τον Απρίλιο συμφωνήσαμε το πρώτο έγγραφο της Προεδρίας. Μετά έγινε μακρά συζήτηση εκ νέου πέντε φορές και στο τέλος όλων αυτών των συζητήσεων και με τη βοήθεια των κρατών μελών που έδωσαν γραπτά σχόλια, εκπονήσαμε την τελευταία εκδοχή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αυτήν που υποβάλαμε και στα κράτη-μέλη. Θα έλεγα ότι στο κείμενο αυτό προσπαθήσαμε να επαληθεύσαμε ένα σωρό πράγματα, αλλά δεν αγγίξαμε τα εκρεμή θέματα που είναι το πεδίο εφαρμογή, οι εξαιρέσει, ε, τα, τα σχέδια επίγουσας δράσης, το ενημέρωση του κοινού κτλ. Θα πρέπει να σας πω ότι στο Συμβούλιο διάφορα κρατημέλη έχουν αποκλίνωσες απόψεις για αυτά τα ζητήματα ε, όσον αφορά δηλαδή το πεδίο εφαρμογή και την ενημέρωση του κοινού. Έχουμε επίσης σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις επιθεωρήσεις. Πιστεύω πως οι εργασίες μας ακολουθούν παρόμοια κατεύθυνση ωστόσο με το Κοινοβούλιο και γι' αυτό και ελπίζω πως η έκβαση θα είναι αίσια. Ελπίζω λοιπόν ότι και στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτή η αγαστή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος από την Κομισιόν που θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις για τις επιθεωρήσεις και για την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας σε Βέζο. Thank ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους όσοι πήραν το λόγο. ιδιαίτερα και τον κύριο Άντερ για την πολύ ε, χρήσιμη έκθεση. Πολλά ζητήματα τα έθηκαν επιτάπητος. Θα ήθελα να πω δύο λόγια καταρχάς για την έκθεση του κυρίου Άντερ. Και στη συνέχεια να ομοδοποιήσουμε κάπως διάφορα θέματα τα οποία ακούστηκαν για να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Για να επανέλθουμε στην έκθεση του κυρίου Άντερ. Καλωσορίζουμε την στήριξη προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα και αυτά που είπε και όσα εξήγησε για το παράρτημα 1, τον τομέα εφαρμογής, στον οποίο πολλοί από εσάς αναφερθήκατε. Χαιρόμαστε που η προσέγγιση μας και σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση του κοινού και την συμμετοχή του κοινού, αλλά και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη, αλλά και τις ε, διατάξεις για τις επιθεωρήσεις υποστηρίχθηκαν στην έκθεση του κυρίου Άντερ. Συμφωνούμε με πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θεωρούμε ότι για κάποιες εξ αυτών θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στη διατύπωση, κάποιες άλλες μας προβληματίζουν λίγο πιο πολύ ως προς τη διατύπωση, αλλά έχουμε και ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί μια παρανόηση. Να το τονίσω, η εισαγωγή προστασίας της ε, περιουσίας αποτέλεσε ένα από τους στόχους το, της οδηγίας. Θεωρούμε ότι δεν είναι ε, δέουσα αυτή η προσθήκη εδώ και ότι θα αύξανε πολύ το πεδίο εφαρμογής. Μπορούμε να το συμπεριλάβουμε μόνο σε ό,τι αφορά την αναφορά ατυχημάτων, όχι υπό την ευρύτερη έννοια. Θεωρούμε δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί γιατί η προστασία της, ανθρώπινα, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος έμεσα περιλαμβάνει και την περιουσία. Επίσης έχουμε κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά το όλο θέμα της παροχής πληροφοριών στο κοινό, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ίσως όμως αυτά να τα κοιτάξω αναομάδες. Αν θέλετε πρόεδρε, να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας για την εφαρμογή, για παράδειγμα. Θα θυμάστε ότι υπάρχει μια έκθεση του Αύγουστου του 2010 που αναφέρει ότι η οδηγία των τελευταίων 15 ετών εφαρμόζεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και οι τομεί όπου υπάρχουν προβλήματα και όπου έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις είναι ο τομέας ακριβώς της πληροφόρησης. Το άρθρο που ρυθμίζει θέματα πληροφόρησης για μέτρα ασφάλειας, για σχέδια πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να διαβιβαστούν με καλύτερο τρόπο προς το ευρύ κοινό. Ένας τομέας λοιπόν, όπου θεωρούμε γιατί και αυτό τέθηκε ως ερώτημα για την εσωτερική οργάνωση των εγκαταστάσεων. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής. Να πω αυτά που είπα και εισαγωγικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα τι κάνουμε, εναρμονίζουμε την ε, οδηγία σε βέζο με αυτά που έχουν συμφωνηθεί, με αυτά που έχουν συζητηθεί στα πλαίσια μια άλλη οδηγία που ανήκει στο πακέτο REACH, την CLP. Και ότι ο λόγος που τροποποιείται η οδηγία σε Βέζο είναι ένας διαφορετικός τρόπος κατάταξης βάσει πιο πολλών πληροφοριών και άλλων διαδικασιών που αποφασίστηκαν στην οδηγία CLP. Άρα ουσιαστικά δεν καθορίζουμε εμείς ε, σε μεγάλο βαθμό το τι γίνεται, γιατί πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις προέρχονται από την οδηγία αυτή. Πολύ σχολιάσατε το θέμα απόκλησης από την ρήτρα α, διασφάλισης. Θεωρούμε ακριβώς ότι προκειμένου να πιάσουμε κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια της οδηγίας σε Βέζο, αλλά περιλαμβάνεται στην οδηγία CLP, συμπεριλάβουμε λοιπόν αυτή τη ρήτρα απόκλησης. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα και σε εθνικό επίπεδο να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από ανεπιθύμητες παρενέργειες της οδηγίας αυτής. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποια ανησυχία για... σε επίπεδο εφαρμογής σε εθνικό, στα εθνικά κρατημέλη και σε ό,τι αφορά και τον ανταγωνισμό, υπάρχουν ανησυχίες. Είμαστε διατεθειμένοι να το ξανακοιτάξουμε αυτό το θέμα από κοινού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούμε ότι προφανώς υπάρχει λόγος να διατηρηθεί αυτή η απόκληση, αλλά ακούσαμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της συναπόφασης, μας είπατε. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να περιμένουμε προκειμένου να εγκριθεί αυτή η νομοθεσία και στη συνέχεια να ελέγξουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε την απόκληση και να περάσουμε σε άλλη συναπόφαση. Άρα επικρατεί η αίσθηση ότι τα κριτήρια θα πρέπει να εφαρμοστούν πρωτού. Τα κριτήρια μάλλον που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την χορήγηση απόκλησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο θα περάσει στην, ε, συναπόφαση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε και ένα εργαστήριο με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη για να σκεφτεί κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο Είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση προς τις πληροφορίες, ανέφερα ήδη ότι ένας από τους λόγους ανησυχίας της τελευταίας έκθεσης ήταν ακριβώς αυτή η ανάγκη για πληροφόρηση. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτά που ζητάμε δεν είναι υπερβολικά. Δεν επισέρχονται σε τομείς όπου θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπερφορτώνουμε το κοινό με υπερβολικές πληροφορίες ή ότι χορηγούμε απόρριτες πληροφορίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν ενδεχόμενε θερμοκρατικές επιθέσεις. Από το κείμενο προκύπτει με σαφήνεια ότι ζητάμε γενικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει τακτικά να ενημερώνονται στο διαδίκτυο, γιατί αυτό αποτελεί το μέσο το οποίο στο οποίο έχουν πρόσβαση πλέον οι πιο πολλοί. Και είναι και το πιο γρήγορο μέσο σε περίπτωση ατυχήματος για τις ενδεχόμενες ουσίες που εμπλέκονται, για τα μέτρα προφύλαξης, για το πώς οι αρχές θα εφαρμόσουν τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την προστασία της υγείας των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν διευκολύνει άλλους στόχους που δεν θα ήταν προς το συμφέρον μας. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις. Όπως ξέρετε, είχαμε συζητήσεις ε, για τις επιθεωρήσεις σε άλλα πλαίσια, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις βιομηχανικές εκπομπές ουσιαστικά η διατύπωση είναι διαφορετική από ότι στην ε, οδηγία για τις ταυτότητες και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ήδη ένας πρώτος έλεγχος ε, κινδύνου τίθενται για απαραίτητε ε, προδιαγραφές με τρόπο που συνάδει με τον τρόπο που έχουμε ακολουθήσει στο παρελθόν. Γιατί άλλωστε να διαφέρει η προσέγγιση μας ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την προσέγγιση που είχαμε στις προηγούμενες οδηγίες. Επιπρόσθετα, φυσικά μπορεί να υπάρχουν επιθεωρήσεις ε, προσδόκητες. Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει προειδοποίηση της διεύθυνσης μιας εγκατάστασης. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, έχω άλλο χρόνο. Ήταν αρκετά συνεκτικά αυτά που είπατε, αναφέρει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά εν Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι δεν ε, υποτιμούμε ενδεχόμενη ανάγκη νομοθετήματος. Αλλά, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, αλλά θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και ελπίζω να σας έπεισα ότι αυτό το θέμα θα το διαπραγματευτούμε, αλλά όχι στα πλαίσια της οδηγίας ΕΒΕΖΟ. Σε ό,τι αφορά τους αγωγούς, θα το εξετάσουμε το ζήτημα και θα δούμε κατά πόσο υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης. Και στο σημείο αυτό θα κλείσω, Πρόεδρε, και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες κατηδίαν. Σας ευχαριστούμε κυρία Βένινγκ για τις απαντήσεις που μας δώσατε να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κάνει τα τελικά του σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έκαναν. Βρίσκομαι στην ευτυχή θέση που μου επιτρέπει να πω ότι ναι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για το θέμα. Είχαμε ήδη πολλές συναντήσεις, οπότε πολλές φορές καταφέραμε να συζητήσουμε με τους θεώδεις εισηγητές όλες τις πλευρές του ζητήματος. Ετέθησαν ορισμένα ερωτήματα, ορισμένες, εκφράστηκαν ορισμένες αμφιβολίες. Το ζήτημα της κοινή γνώμη, πιστεύω θα είναι ένα από τα πιο αντιμεχόμενα σημεία. Αν κρατήσουμε το κείμενο έτσι όπως μας το εξήγησε η κυρία Βένινγκ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η Κομισιόν το είπε. Θέλει να βάλει γενικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας το ανέφερα. Πληροφορίες για τους περίκους να εξηγούν ποιες είναι οι επικίνδυνες ουσίες που περιτριγυρίζουν τον κοσμάκι, να δίνονται οδηγίες, τι συμπεριφορά πρέπει να κρατήσουν οι κάτοικοι σε περίπτωση καταστροφής. Αυτό αδιαμφισβήτητα. Το πρόβλημα όμως υφίσταται αν φυσικά περάσει η πρόταση της Κομισιόν, ότι θα καταλήξουν στο διαδίκτυο και ένα σωρό τεχνικές πληροφορίες, κατάλογοι, μητρώα. Αυτό δεν είναι χρήσιμο, δεν βελτιώνει την ασφάλεια. Ίσα ίσα θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση στους πολίτες. Όπως ε, και τα πρακτικά του ελέγχου. Αν κάτι τέτοιο δημοσιευόταν στο ίντερνετ, ο ενδυνάμει τρομοκράτης κάλλιστα θα μπορούσε να πάει στο ίντερνετ για να δει ποια είναι τα αδύνατα σημεία του εργοστασίου και να κάνει τη δουλειά του. Γιατί λοιπόν εμείς να δημιουργήσουμε δυσχέρειες ε, στην, στα ζητήματα ασφάλειας και να ενισχύουμε και τους ενδυνάμει τρομοκράτες. Τώρα, Αν υπάρχει παρερμηνία, τότε μπορούμε κάλλιστα να τροποποιήσουμε το κείμενο και να τελειώνει υπόθεση. Για το φαινόμενο ντομινό που ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι για τις παρεμβολές με άλλα εργοστάσια, κοντινά εργοστάσια. για να συνεννοούμεθα. Αν έχουμε δύο χημικά εργοστάσια, το ένα κοντά στο άλλο, η Κομισιόνα ε, για, για το νέο εργοστάσιο το οποίο έρχεται να εγκατασταθεί στο, δίπλα σε κάποιο άλλο εργοστάσιο, κοντά σε ένα άλλο εργοστάσιο, να ζητήσει όλες τις πληροφορίες και να τις έχει. Διότι άμα αυτή η καινούργια επιχείρηση, το καινούργιο εργοστάσιο που πάει να φτιαχτεί κοντά στο παλιό δεν έχει πληροφορίες, δεν μπορεί να αναλάβει κανείς την επένδυση. Και βέβαια οι πληροφορίες στην τροπολογία 21 είναι αυτά. Ε, πρέπει να δίνονται τα τάχιστα για να μπορεί ο, ο, ο επιχειρηματίας να επενδύει γρήγορα. Μετά έχουμε και τον συνάδελφο Κράμερ, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε μεγάλες χημικοί μεγάλα χημικά εργοστάσια στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά ο, με τη νέα... Με, την νέα οδηγία, με, με την τροποποίηση, τότε θα έχουμε αύξηση. των εργοστασίων στην περιοχή του. Αν τώρα ο συνάδελφος Κράμερ έχει αποδείξεις που λένε σαφές, σαφώς ότι μετά από την έγκριση αυτής της ρύθμισης θα αυξηθεί κατά 30% ο αριθμός των μονάδων που θα ενταχθούν στο εφαρμοστικό πεδίο να μου το πει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Άντερ. Ο κύριος Κράμερ θα σας ε, δώσει τους υπολογισμούς αυτούς που καταλήγουν σε ποσοστό 30% και όχι 10% και να δούμε κατά πόσον θέλουμε μια τέτοια ε, αύξηση. Μάλιστα. Ήταν λοιπόν καρποφόρα η συζήτηση. Προθεσμία καταθέση τροπολογιών είναι 23 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο ε, στην Επιτροπή μας και το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια η έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και περνάμε στο 4 της ημερής διάταξης προστασία των αποθεμάτων πόσιμου είδατος. Μας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προβλέπεται Μα δεν είναι απαραίτητη τροποποίηση της νομοθεσίας, αλλά φυσικά μας αφορά το θέμα αυτό ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θέλουμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία αυτή για το θέμα αυτό. Ε, καλέσαμε λοιπόν την Κομισιόν να μας παρουσιάσει το θέμα ο κύριος Μπλούς από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα μας χορηγήσει τις πληροφορίες αυτές. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the Commission is grateful for this invitation. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή είναι ευγνώμων για την πρόσκληση αυτή ε, που έγινε μετά από την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ ημών, κύριε Πρόεδρε, και του Επιτρόπου Τόμσκιν. Ναι. Εμείς έχουμε εξετάσει το θέμα του πόσιμου ύδατος από διάφορες οπτικές γωνίες. Από τη μια πλευρά εξετάσαμε την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζεται με το πόσιμο ύδατος. Από την άλλη πλευρά, εξετάζοντας το, ποιότητα του πόσιμου ύδατος στην βρύση του καταναλωτή και προστασία των αποθεμάτων ε, πόσιμου ύδατος καθώς και του περιβάλλοντος όσον αφορά την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα. Θα ξεκινήσω, Πρόεδρε, με την εγκυρότητα των παραμέτρων και των αξιών που θεσπίζονται από την Οδηγία Πόσιμου Ήδατος. Το πόρισμα της Επιτροπής αυτή την χρονική στιγμή είναι ότι οι παράμετροι και οι αξίες και οι τιμές μάλλον εν γέννη αντικατοπτρίζουν τις διαθέσιμες γνώσεις ε, και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναθεώρηση των παραμέτρων και των τιμών, πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο με την ε, συνήθη διαδικασία. Ωστόσο, η Κομισιόν θα συνεχίσει να εξετάζει προσεκτικά τις επιστημονικές εξελίξεις όταν αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να προτείνει αναθεώρηση όταν θα χρειαστεί. Ταυτόχρονα, ορισμένε τεχνικέ ε, λεπτομέρειε για την δειγματοληψία και ανάλυση του πόσιμου είδου χρειάζονται ενημέρωση ε, και έτσι, όπω ε, την υποχρεώνει η οδηγία, η Κομισιόν θα θα κάνει αυτή την ενημέρωση σύμφωνα με την συνηθισμένη διαδικασία ε, εξέτασης της πρότασης αυτής. Τώρα, για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος στο βρύση του καταναλωτή γεν γέννη υπάρχει μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης για τις μεγάλες ε, παροχές νερού που εξυπηρετούν πάνω από 5.000 ανθρώπους δηλαδή. Η συμμόρφωση είναι πάνω από 80%. Ωστόσο, σε μερικές περιοχές η συμμόρφωση για μικρές ε, παροχές, για την εξυπηρέτηση 50 και 5.000 ε, πολιτών υπάρχουν προβλήματα με 30 ίσως και 40% της παροχής μη συμμορφούμενο προς τις ε, διατάξεις. Όπως ε, αναφέρθηκε στην επιστολή του Επιτρόπου ποδέώ είναι και η Κομισιόν έχει προτείνει μια πολλαπλή προσέγγιση. Από μια πλευρά, ανάπτυξη καλών πρακτικών και γράφου για τις καλύτερες πρακτικές επί τη βάση των εμπειριών των κρατών μελών, προώθηση της εκτίμηση κινδύνου για τις μικρές παροχές και από την άλλη πλευρά ε, μέτρα επιβολής επί τη βάση της υποχρέωσης συνεργασίας που εγγράφεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις παροχές που δεν έχουν υποχρέωση να αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο ή στην Επιτροπή. Τέτοια αιτήματα για τα στοιχεία έχουν ήδη εκδοθεί και έχουν δοθεί στα κράτη-μέλη και διμερός θα έχουμε επαφές με τα κρατη αλλά και, θα αναλάβουμε δράση επιβολής υπό τα άρθρα 208 και 16, 216 της συνθήκης, αν χρειαστεί. Τώρα, προστασία του πόσιμου ύδατος και του περιβάλλοντος για να σας θυμίσουμε το η ναυαρχίδα της οδηγίας πλαισίου περί πόσιμου ύδατος. με στόχος ήταν να έχουμε καλύτερο πόσιμο ύδωρο και καταρχήν θεσπίζεται υποχρέωση για προστασία των υδάτων. Επίσης και για την αφαλάτωση του παράκτηου ύδατος ε, προβλέπονται ειδικέ προδιαγραφές ποιότητας αλλά και ειδική προστασία για τα ύδατα που χρησιμοποιούνται ως πόσιμα, πόσιμο ύδερο ή σκοπεύουν να χρησιμοποιηθούν ε, ως τέτοιο στο μέλλον. Τα περισσότερα κρατημέλη έχουν θεσπίσει προγράμματα και σχέδια ε, μέσα στις προθεσμίες. Μάλιστα, τέσσερα τέσσερα κράτη-μέλη έχουν ήδη παραπεμφθεί στο, δικαστήρι, στο 10, Πορτογαλία, η Ελλάδα, η, η Γερμανία και το Βέλγιο και από ό,τι φαίνεται ήδη έχει εκδοθεί γνωμοδότηση για την Ισπανία. Για το μέλλον, ξέρετε ότι ο Επίτροπος Ποτόσνικ έχει δεσμευθεί να υποβάλει πριν το πέρας του 2012 προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια πρόταση για προστασία του κόσμου είδου της Ευρώπης που θα παρουσιάζει καταρχήν μια αξιολόγηση της Επιτροπής για όλα τα σχέδια και προγράμματα υπό την οδηγία πλαίσιο για το πόσιμο νερό. Εμείς είμαστε γνώμενες στο Κοινοβούλιο διότι δώσατε σημαντικά κονδύλια για πιλωτικά προγράμματα αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων Έπειτα ε, θα εξετάσουμε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις ε, για την λειψιδρία και την ξηρασία. Κάτι που αφορά όχι μόνο τα νότια κράτη-μέλη, αλλά και άλλες ε, χώρες που μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όσον αφορά την, τον ανεφοδιασμό νερού και έπειτα συμπεράσματα και προτάσεις για την οδηγία για το περιβάλλον και το νερό και όλα αυτά βέβαια, βεβαίως μέσα σε πλαίσιο διαφάνειας, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ, την επιστημονική κοινότητα και τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται και φυσικά οι, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα θα δημοσιευθούν και στο ίντερνετ. Εμείς προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας μέσω της, ε, του Intergroup για το νερό, το οποίο προεδρεύει ο κ. Σέμπερ, που είναι και μέλος αυτής της Επιτροπής. Να θυμίσω ότι η προστασία των ε, υδάτινων πόρων μας θα χρειαστεί διαρκώς επενδύσεις ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερη σημασία όταν αποφασίζουμε για τα επόμενα προγράμματα. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομο, κύριε Πρόεδρε, και προβλέπω και είμαι διαθέσιμος για να απαντήσω σε ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή στη συζήτηση. Το πόσιμο είδωρ αποτελεί το πρώτο αγαθό για την επιβίωση. Αυτό πάντα το επαναλαμβάνουμε και φυσικά προστασία του πόσιμου είδατος αποτελεί ε, ζωτική σημασία σε ανάγκη. Μας αναφέρατε τις παραμέτρους και τις τιμές που ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες ε, τεχνολογίες και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή επί του παρόντος για τη λειψιδρία που αποτελεί ένα σημαντικό θέμα τουλάχιστον για την Νότια Ευρώπη. Αυτή τη χρονιά αποτέλεσε θέμα και αποτελεί θέμα και για την Κεντρική Ευρώπη έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό και ακόμα και βόρεια των Άλπαιων η κατάσταση νομίζω θα καταστεί αρκετά δύσκολη. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια ενιαία, ένα ενιαίο σχέδιο για την κλειψιδρία ε, και για την εξοικονόμηση νερού και ίσως να υπάρχουν διαφοροποίησεις, γιατί ίσως να υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλα πρόβλημα λευσιδρέας. Δεν έχει λοιπόν νόημα και αυτή η επιβολή προορισμών. Μία ερώτηση η οποία πάντα ακούγεται στη Γερμανία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού αποτελεί θέμα των δημοτικών αρχών. Κάθε δήμος ε, είναι αρμόδιος για το πόσιμο νερό. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά προωθεί την ενιαία αγορά, την απορρίθμιση δηλαδή. Εσείς ε, θεωρείτε ότι αποτελεί τομέα αρμοδιότητά σας? Αναφέρετε στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές ε, συμβάσεις. Εδώ οι απόψεις δίστανται για το κατά πόσον ε, αυτό θα ήταν προ όφελο τη ποιότητα. Είναι ήδη υψηλή η ποιότητα, ίσως δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να κάνετε κάποια σχόλια. Ο Βιτόριο Πρώτη, που ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την τοποθέτησή της με την οποία βεβαίως συμφωνώ αλλά επιφυλάσσομαι μόνο σε μερικές λεπτομέρειες διότι εμείς τίνουμε προς μία σημαντική αλλαγή του πλαισίου των βροχοπτώσεων και έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές που είναι πλέον πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι χρειάζεται μία πολιτική πιο γενική και πιο αποτελεσματική για τη διαχείριση του ύδατος παράλληλα με την διατήρηση της ε, επικράτειας διότι το κλίμα έχει αλλάξει. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως θα έπρεπε να έχουμε και μία επαναδιοχέτευση, μία ένεση υδάτων στα υπόγεια φρεάτια ούτως ώστε να τα τροφοδοτήσουμε στα αποθέματά τους, τα οποία είναι αποθέματα πόσιμου νερού. Επίσης, λέγαμε για τους Δήμους να υπάρξει μία ειδική δράση έναντι της αδιαφροχοποίησης του εδάφους σε αστικό περιβάλλον. Να μπορέσουμε λοιπόν και στα υπόγεια αστικά φρεάτια να σε αυτά τα φρεάτια λοιπόν να διοχετεύσουμε εμείς απ' έξω νερό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επαρκή αποθέματα. Πρέπει να επανεξετάσουμε επίσης και τη γενική πολιτική για το νερό την οδηγία πλαίσιο για το νερό και αυτό πάντοτε σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Είναι υπεραπαραίτητο να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να βελτιώσουμε και την ποιότητα του νερού αλλά και να μας δοθεί δυνατότητα της δημιουργίας αποθεμάτων, ε, νέων υδατικών αποθεμάτων και προστασίας των υπογείων φρεατίων. Η Λίντα Εύανς. Δεν άκουσα, δεν άκουσα την αρχή της παρέμβασής σας, γι' αυτό συγχωρέστε με. Αντί να φτιάξετε νέα νομοθεσία, λέτε για οδηγό καλύτερης πρακτικής, καλύτερων πρακτικών. Με ποιο στόχο, ποιο θα είναι ο στόχο σα και τι κάνετε με τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική, ποια είναι η εμπλοκή σα σε αυτά. Εγώ την Παρασκευή ήμουνα ε, έξω στο Yorkshire, ήταν μια, σε μια πολύ κρύα και βροχερή μέρα στο Yorkshire και κοιτούσα τι επιπτώσει τη διάβρωση ε, το στο πόσιμο νερό. Το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι είναι ότι δεν έχουν ε, την γη, οι γεωργοί έχουν αυτή την ε, γη και αυτοί που έχουν ε, τη γη για να κάνουν κάποια, αθλητικο, κάποια αθλήματα. Και φυσικά υπάρχουν και οι εταιρείε διανομής του νερού. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι ο φορολογούμενος είναι αυτός που πρέπει να πληρώσει. Αν για παράδειγμα εσύ αποφασίσεις να καθαρίσεις την ε, έλλη και την τύρφη, ναι, κερδίζεις από την τύρφη, αλλά αντίθετα επιβαρύνεις την ποιότητα του νερού και ο φορολογούμενος είναι αυτός που θα πληρώσει να καθαρίσει το νερό και να ξαναποκτήσει την κανονική του ποιότητα. Τώρα έχουμε μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, μπορούμε να ξαναδούμε τις πρακτικές ε, της γεωργίας για τη διαχείριση των γεών, την χωροταξία. Εσείς ασχολείστε με αυτό. Μπορείτε να ασχοληθείτε μειώνοντας τα όσα φτάνουν στον πόσιμο νερό και επιτά. μήπως πρέπει να διατηρηθούν αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά, και είναι και οικονομικό το θέμα για τους φορολογούμενες ε, Φυσικά χαρακτηριστικά όπως τα έλλη τύρφη. Κρίστα ευχαριστώ το νερό αποτελεί ένα διαρκές ε, θέμα που μας απασχολεί και μιλάμε σήμερα για τα αποθέματα πόσιμου νερού. Θα ήθελα να θέσω λοιπόν δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυρία Πλούς. Μιλάμε για εξοικονόμηση πόσιμου νερού για τη διατήρηση των αποθεμάτων. Ίσχυει ότι σε κάποια ε, μέρη της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης ε, η υπερβολική εξοικονόμηση νερού προκαλεί και αυτή προβλήματα γιατί για παράδειγμα ε, βρωμίζουν οι αγωγοί γιατί δεν περνάει αρκετό νερό και πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά που προκύπτουν είπε ο πρόεδρος Γιολάιν ότι είναι διαφορετική η πρόσβαση στο νερό σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να είναι διαφορετική η προσέγγισή μας. Επιπλέον, αύριο θα ψηφίσουμε την οδηγία για τα απορριπαντικά. Θα απαγορεύσουμε το... διάφορες ουσίες στα απορριπαντικά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον ειδικό για θέματα νερού κατά πόσο αυτό είναι καθοριστικό για το πόσιμο νερό για το κατά πόσον θα απαγορευτούν οι ουσίες αυτές ε, και σε ό,τι αφορά τα απορριπαντικά για τα πιάτα ή κατά πόσο θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ κύριε Ντέιβις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Βικτώριο Πρόντι. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ την ανάγκη ένεσης νερού στις, ε, στα φρέαδια κατά από τις πόλεις για ε, αποτραπούν ε, ενδεχόμενες αποσταθροποίησεις. Αλλά ξέρω ότι στο Μεξικό είναι τεράστια τεράστιες ποσότητες αυτές. Δεν έχω δει στατιστικά στοιχεία, ωστόσο, ούτε για τις ευρωπαϊκές πόλεις. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει νόημα να υπάρξει νέα νομοθεσία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο υπάρχει νομοθεσία η οποία ακόμα δεν έχει σωστά εφαρμοστεί από τα κρατημέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε κάποιες δράσεις που έχουν αναλυφθεί για την εφαρμογή σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, αλλά και σε ό,τι αφορά την Ισπανία και τη Σλοβενία ενδεχομένω, αλλά αυτό σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Από ό,τι άκουσα, ο Επίτροπος έχει δεσμευτεί απέναντι στην Επιτροπή μας να προσπαθήσει να εφαρμόσει την νομοθεσία με το δέοντα τρόπο και να καταστεί αυτό υψηλή προτεραιότητα. Αλλά έχω την αίσθηση ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ε, κατά των κρατών μελών για να πετύχει την σωστή εφαρμογή. Μπορούμε να έχουμε και πολλές πληροφορίες και για τα βήματα που γίνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μελη θα κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν να κάνουν. Ευχαριστώ και τελευταίος ο κύριος Στοδαριλα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν εμείς υποστηρίζουμε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της έλλειψης νερού, αναρωτιέμαι γιατί το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέχουν ιδιαίτερα τις κλιματικές αλλαγές και όχι τόσο την έλλειψη του ύδατος. Εγώ εύχομαι για αυτό το θέμα του νερού τόσο η Κομισιόν όσο και το Κοινοβούλιο να αρχίσουν να προσδίδουν την απαραίτητη προσοχή διότι εμείς ε, μπορούμε κάλλιστα να συνεχίσουμε να ζούμε σε έναν κόσμο με μολυσμένη ατμόσφαιρα αλλά σε έναν κόσμο χωρίς νερό μπορεί να προκύψουν πόλεμοι και να πεθάνουμε. Εγώ δεν διαπιστώνω να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της εξοικονόμησης του νερού. Φτάνει κανείς να σκεφτεί ότι στο Τάραντο η μεγαλύτερη Ιταλική χαλιβουργία τροφοδοτείται με πόσιμο νερό. Αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος τροφοδότησης του χαλιβουργίου της Ήλβα. Από το πρωί, στην καθημερινή μας ζωή, όταν πλένουμε τα δόντια μας και σε όλη την ημέρα, πόσο νερό καταναλώνουμε που θα μπορούσαμε να το είχαμε εξοικονομήσει και αυτό καθιστώντας υποχρεωτικά ορισμένα μέτρα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, αισθητήρε λοιπόν για να μπορούν να διαπιστώνουν πότε έχουμε διαφυγή νερού και να μπορούμε να εξοικονομούμε. Και μετά σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του και το θέμα της εξοικονόμησης του νερού. Μιλάμε εμεί για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Δεν θα έπρεπε να προβληματιστούμε προς τις καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν λιγότερο νερό, αλλάζοντας την τυπολογία δηλαδή της καλλιέργειας να εξοικονομήσουμε εκατομμύρια λίτρα νερού το ενδιαφέρον εμένα πάντως σήμερα μου φαίνεται λίγο περιορισμένο. Κύριε Βλέσσα, άκουσα ότι είπαν οι συνάδελφοι. Σας παρακαλούμε λοιπόν να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με το δικό σας το ερώτημα σε ό,τι αφορά τα θέματα οργάνωσης για την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων, το οποίο γίνεται βασικά από τα Δημοτικά Συμβούλια στη χώρα σας να επαναπιβεβαιώσω το εξή. Το θέμα το πώς κάθε χώρα βάσει του συντάγματός της οργανώνει την παροχή δημόσιου ύδατος μέσω ιδιωτικών ε, ε, εταιριών, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι θέμα των περιφερειών. Το 345 άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητά απαγορεύει οποιαδήποτε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην νομοθεσία που αφορά τα θέματα ιδιοκτησίας ε, στις ε, χώρες μέλη. Έγινε και ένα σημαντικό δημοψήφισμα στην Ιταλία πρόσφατα όπου τέθηκε το ερώτημα στο εκλογικό κοινό κατά πόσο θα ήταν υπέρ της ιδιωτικοποίησης της παροχής ε, της συντροδότησης. Αυτό είναι κάτι το θεμητό το οποίο μπορούν να τα συζητούν τα αρμόδια σώματα στην Ιταλία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όχι όμως οι Βρυξέλλες. Δεύτερο στοιχείο στο πλαίσιο αυτό είναι τα θέματα δημοσίων προμηθειών. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα της ιστορικής ανάθεσης συμβάσεων ή της εξωτερικής ανάθεσης, outsourcing. Ένα παράδειγμα να δώσω για όσους δεν ε, γνωρίζουν απαραίτητα την κατάσταση. Αν στην Βιέννη δημιουργούταν μια εταιρεία 95% στα χέρια του Δήμου της Βιέννης και 5% στα χέρια του κρυού Μπλεχ, του φαινόμενου και μετά ετήφετο τη σύμβαση στην εταιρεία αυτή για την υδροδότηση με πόσιμο νερό. Το δικαστήριο έχει αποφανθεί στο παρελθόν ότι το 5% του κυρίου Μπλουχ και το 95% για το Δήμο της Βιέννης αποτελεί σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικό τομέα και άρα υπόκειται στους κανόνες και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που φυσικά αυτό δεν θα ωφελούσε το Δήμο της Βιέννης, γιατί θα έπρεπε να έχει προσωπικό χιλιάδων ε, ατόμων για την ε, λειτουργία της εταιρεία και παρόλα αυτά να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Αλλά είναι σαφείς οι κανόνες πλέον. Και στο πλαίσιο αυτό η ευθύνη είναι στα χέρια των ε, κρατών και των περιφερειών, προκειμένου να επιλέξουν την καλύτερη κατάσταση για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες αυτές και οι παραδόσεις είναι διαφορετικές. Τρεις τύπους έχουμε ουσιαστικά χονδροειδώς στην Ευρώπη. Οι Δήμοι, τα Δημοτικά Συμβούλια, που ε, ρυθμίζουν θέματα υδροδότησης με πόσιμο νερό. Δεύτερο μοντέλο ιδιοκτησία στους Δήμους, αλλά η καθημερινή διαχείριση ε, έχει ανατεθεί εξωτερικά σε παρόχους και τρίτο μοντέλο, το οποίο επικρατεί μόνο στην Αγγλία και στην Ουαλία, όχι στη Σκοτία, όχι στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου είναι δημόσια ιδιοκτησία στα δίκτυα ιδρυδότηση. Στην Αγγλία λοιπόν και στην Ουαλία έχουμε ιδιωτικέ επιχειρήσει και για την ιδιοκτησία αλλά και για την καθημερινή διαχείριση. Στο ερώτημα του κυρίου Πρόντι για την ε, εκ νέου χρήση του ύδατος υποστηρίζω πολύ τι θέσει που υποστηρίζει αυτή η εκ νέου αξιοποίηση θα αποτελέσει ένα μεγάλο, μια μεγάλη απάντηση στη λειψιδρία για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση για την ε, ξηρασία και για τη λειψιδρία ανέφερε τέτοιε λύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Κύπρος είναι πολιτική της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου ότι ο στόχος είναι 100% επαναχρήση του νερού. Να μην ε, χύνεται ούτε ένα κυβικό μέτρο νερού στην Μεσόγειο. Να χρησιμοποιείται για την άρδρευση, για τη γεωργία. Και να σας πω ότι Όλοι, όλα τα σύνορα της ε, Κύπρου είναι στις ακτές, άρα έχουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Να αναφερθώ στον κύριο Ντέιβις τώρα. Οι δραστηριότητες οι βιομηχανικές και οι αγροτικές έχουν οδηγήσει σε υψηλές ε, τιμές, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη χρήση των ε, υπόγειων υδάτων, αλλά έχει να κάνει και με θέματα διάβρωσης και πλημμύρων. Όπου είναι δυνατόν λοιπόν, να προσπαθούν, ε, όπου είναι δυνατόν προσπαθούμε να διοχετεύσουμε το νερό της βροχής στο έδαφος. Αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντέιβιτ, προαπαιτεί κάποια νομοθεσία, αποτελεί βέλτιστη πρακτική, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα της οδηγίας για το πλαίσιο του νερού τρίτο τμήμα. Δυνατότητα εξοικονόμησης νερού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει δύο βασικές πηγές όπου μπορεί να γίνει εξοικονόμηση νερού. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά η άρδευση για τη γεωργία, που σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στο νότο όπου υπάρχει η λειψιδρία, συμβάλλει, μάλλον αντιπροσωπεύει σε 85%, 85 της χρήσης νερού. Και κατά δεύτερον, διαρροές. Υπάρχουν, και υπάρχουν ακόμα ε, εκατονταετή συστήματα εδροδότησης με μεγάλες διαρροές. 50%. Άρα αυτές οι διαρροές ε, θα πρέπει να διορθωθούν και αυτό θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού. Ο κύριος Λάινεν εξέφρασε κάποιες ανησυχίες. Να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ να καταθέσει μία ενιαία πρόταση ανεξάρτητα από το τι διαρροές υπάρχουν 1%, 2% ή 60-70% θα πρέπει πάντα να προσαρμόζονται αυτές οι νομοθεσίες στις ανάγκες της περιοχής. Για την κυρία Μακέβαν να πω το εξή το έγγραφο για τις βέλτιστες πρακτικές θα διατεθεί κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο ήμιση του 2012 και στόχο θα έχει ακριβώς αυτές τις προμήθειες νερού, την παροχή νερού, ε, όπου υπάρχουν σήμερα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία είναι η γεωλογική μόλυνση σε μεγάλο βαθμό μετά από τα περιστατικά, με τα αγκούρια, με τα Όλοι ξέρετε τα περιστατικά με, στη Γερμανία και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με μη συμμόρφωση σε μικρές ε, γεωργικές καλλιεργίες. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις συγκεκριμένες περιοχές ε, Παροχή νερού όπου υπάρχουν προβλήματα και μαζί με τα κρατημέλη και με τις δήμους αυτούς θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Πολύ επίκαιρο και εύστοχο ερώτημα. Ο Επιτροπός μου είναι απόλυτα δεσμευμένος για την πολλαπλή συμμόρφωση με την οδηγία για το πλαίσιο για το νερό στο, πλε... στο... στη μελλοντική διαμόρφωση της ΚΑΠ ως ε, προαπαιτούμενο για επιχορηγήσεις. Γιατί πλέον ισχύουν και το κοινό και οι γεωργοί ξέρουν, ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται να κάνουν προκειμένου να συμμορφώνονται. Αυτό πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν έτσι. αναφέρθηκαν ήδη στο ότι σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση νερού, ποτέ δεν θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ενιαία λύση που θα ταιριάζει σε όλους. Άρα η ερώτηση της κυρίας Κλάς νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε πάντα μία λύση η οποία θα ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε περιοχής και όχι να λύσουμε ένα πρόβλημα ε, δημιουργώντα ένα άλλο κατά δεύτερον, τέλος μάλλον, σε ό,τι αφορά τα φωσφορικά άλατα και τα απορριπαντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει μια πρόταση μέχρι το 2015 για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι στο κοινοβούλιο αυτό εξετάζεται διάφορες ιδέες και ότι δεν ήταν δυνατό να ληφθεί μία απόφαση για την κατάργηση και το φωσφορικό άλατος στα απορριπαντικά για τα πιάτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η απόφαση της επηρεάζει διάφορες χώρες, 16 χώρες των ΙΠΑ έχουν ήδη λάβει νομική, αναλάβει νομική δράση για την κατάργηση του φωσφορικού άλατος από την ε, βιομηχανία, από τον κλάδο, οι απαντήσεις είναι διτές. αυτό εξαρτάται και με το ποιον μιλάει κανείς. Αλλά είμαι βέβαιος ότι η πολιτική διαδικασία θα καταλήξει στην εξέβρεση μιας λύσης και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν μια τέτοια λύση. Ο κύριος Ντέιβις έθεσε μια ερώτηση για το κατά πόσον είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσια για το νερό. Η απάντηση των περιβαλλοντολόγων θα ήταν ότι πάντα μπορεί κανείς να είναι πιο φιλόδοξος, αλλά κοιτώντα ε, το χρονοδιάγραμμα, το 2010, το Μάρτιο, ε, έκανε σχετική ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο μήνες μετά ξεκίνησε διαδικασία παραβάση και λιγότερο από ένα χρόνο μετά ξεκίνησε την πρώτη από τις έξι ε, αγωγές προς τα δικαστήρια. Η εικόνα λοιπόν 21 χωρών που ακολουθούν το πρόγραμμα καταδεικνύει ότι η στρατηγική εφαρμογής που καταρτίστηκε από τα κρατημέλη, από τις περιφέρειες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς απέφερε καρπούς. Όσοι δεν έκαναν ε, τη δουλειά τους θα παραπεμφθούν στο δικαστήριο φυσικά. Τέλος, Πρόεδρε, για αυτό που είπε ο κύριος Ταταρέλα. Ναι, αναμφίβολα η αλλαγή του κλίματος αποτελεί ένα βασικό κινητήριο μηχανισμό για την διαχείριση των υδάτων. Και ίσως η τρέχουσα ξηρασία στην κεντρική και δυτική Ευρώπη θα υπογραμμίσει την ανάγκη ανάληψης δράσεων. Αλλάζει το ποσοστό βροχοπτώσεων και αυτό επειδή η μέση βροχόπτωση ανά έτος παραμένει λίγο πολύ η ίδια, προκαλούνται και πλημμύρες. Και αυτό θα αλλάξει τα στοιχεία υδρογραφίας σε ό,τι αφορά και τις πλημμύρες θα αλλάξει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τόσο τελεχώς συλλέγανε οι προηγούμενες ε, γενιές. Μια κουλτούρα εξοικονόμησης νερού θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ζωής μας, όχι όμως ε, μόνο στα νοικοκυριά, σε ό,τι αφορά τα καζανάκια, τα ντους κτλ, αλλά κοιτώντα και τους μεγάλους καταναλωτές τους οποίους ε, ε, εξήγησα ήδη ποιοι είναι, η γεωργία και οι απώλειες σε μεγάλα δίκτυα υδροδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πλούς για τις απαντήσεις αυτές που μας δώσατε. Το θέμα θα συζητηθεί σίγουρα σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και περνάμε σε δύο σημεία α, ακόμη πρωτού έρθει στις 5.30 ο κύριος Ντάλι. Έχουμε 15 λοιπόν λεπτά για δύο θέματα. Περνάμε στο 5 τροποποίηση της οδηγίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των φάσεων εκπομπών στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο. Ο κύριος Ταταρέλα είναι ο ειδικός μας. Θα είμαι τηλεγραφικός πρόεδρε, διότι αυτή η Επιτροπή ήδη δύο φορές ασχολήθηκε με το θέμα σε μία δική μου έκθεση και σε μία έκθεση της κυρίας Πιτικάνεν. Και αυτή η έκθεση αποτελεί τη συνέχεια του όλου πλησίου. Διότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πάντοτε το ίδιο. Θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης ε, εκτίμησε ότι θα πρέπει να περιορίζονται σταδιακά και όρισε διάφορες χρονικές φάσεις. Στις άλλες δύο σχέσεις, ε, εκθέσεις ασχοληθήκαμε να αυξήσουμε την ελαστικότητα που δώσαμε στον νομοθέτη. Εδώ όμως δεν θέλουμε να αυξήσουμε την ευελιξία, την ελαστικότητα. Θέλουμε να καταργήσουμε την οδηγία. Τουλάχιστον τη φάση 3β και 4. Και αυτό για έναν απλούστατο λόγο. Ασχολούμαστε. Αυτό αφορά σε ελκυστήρες πάρα πολύ μικρούς. Δηλαδή με μικρό μετατρόχιο. Σχεδόν παιχνιδάκια. Το, φάρτο το μεγαλύτερο τέτοιο τρακτέρ κατασκευάζεται στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη. Τώρα, το σύστημα του ελκυστήρα είναι αρκετά ογκώδες και δεν μπόρεσε να βρει η τεχνολογία ένα τέτοιο σύστημα που να μπορέσει να ένταχθει στα πλαίσια μέσα στους ε, στις ε, μηχανές ή στο σασί. Τεχνικά λοιπόν κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Η στο δε πρότεινε αυτή η τρίτη και η τέταρτη φάση να μην εφαρμοστούν σε αυτού του τύπου τους ελκυστήρες. Η Κομισιόν βρήκε μια σολομονική λύση με την οποία συμφωνώ. Δηλαδή για τρία χρόνια να στέλνει την ισχύ αυτού του μέτρου. Δηλαδή τις φάσεις 3 και τις φάσεις α για να, λέει για να μπορέσει να προσαρμοστεί η βιομηχανία. Αυτό είναι βέβαια, ξέρετε, δύσκολο και χρειάζεται το 2014 να γίνει μία επαλήθευση για να δούμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση ή να το παρατήσουμε εντελώς αυτό το μέτρο. Ευχαριστώ κύριε Δευταρέλα. Σύντομος και περιεκτικός. Σαφέστατος. Προτείνεται λοιπόν να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ε, αναβάλουμε την εφαρμογή της φάσης 3 και 4 κατά τρία χρόνια και να δούμε κατά πόσο θα βρεθούν λύσεις. Η κυρία Κράμα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ο κύριος Κράμα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πάντα φαίνεται ότι θεωρούμε ότι είναι του διαβόλου να αναβάλουμε μια ισχύουσα νομοθεσία και αυτό αντανακλαστικά θα προκαλέσει αντιδράσεις από τους πράσινους. Να προσέξουμε σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ε, επιβλαβών ουσιών να μην ε, εξαιρέσουμε την νεοκυλίνη. Βελτιώσαμε κάποια στοιχεία. Γράψαμε κάτι επιθυμητό στην νομοθεσία. Και στη τελική ανάλυση αυτό δεν εφαρμόζεται. Είπε ο κύριος Τοταρέλα ότι πλέον ένα μικροσκοπικό κομμάτι της αγοράς αφορά αυτά τα μικρά τρακτέρ. Και η παραγωγή των τρακτέρ αυτών μας έρχονται και μου λένε ότι υπάρχουν ήδη όρια εκπομπών και στο επόμενο βήμα θα αποκτήσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί προαπαιτεί τεχνολογίες οι οποίες είναι μεν διαθέσιμες αλλά δεν υπάρχει χώρος κατασκευής σε αυτά τα μικρά τρακτέρ. Και αυτό το καταλαβαίνω γιατί βλέπω ότι για παράδειγμα στα μεγάλα φορτηγά υπάρχουν όρια για τις επιβλαβείς εκπομπές Και αυτή η μείωση των εκπομπών είναι εξίσου ογκώδης και εξίσου ακριβή όσο και ο ίδιος ο κινητήρας. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι για το μερίδιο της αγοράς που μιλάμε δεν ξέρω πόσα τρακτέρ κατασκευάζονται στην Ευρώπη, δεν είναι πάρα πολύ. Οι εκπομπές και τα πρότυπα που ισχύουν δεν είναι μετρήσιμα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό που συζητάμε. Μιλάμε για λιγότερο από 1%, πολύ λιγότερο. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε στο σημείο αυτό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σας πω ότι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό γιατί είναι προβλέψιμο και σε τρία χρόνια όταν θα τεθεί σε εφαρμογή νομοθεσία αυτή δεν θα έχει μεγεθυνθεί ο χώρος ε, κατασκευής σε αυτά τα μικρά τρακτέρ και να σας υπενθυμίσω ότι θα κλαίμε αν δεν μπορούμε πλέον να κατασκευάζουμε τέτοια μικρά τρακτέρ γιατί θα καταστεί αυτό τεχνικώς αδύνατον από τις τεχνικές προδιαγραφές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Η ελπίδα φυσικά υπάρχει ότι θα υπάρχουν καλύτερες τεχνικές ε, λύσεις. Ο κύριος Άικοτ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Εγώ πριν φύγει, πριν φύγετε, σας έχω μια καλή έκπληξη. Εμείς πάντα κοιτάμε το περιεχόμενο και μετά αποφασίζουμε τι να κάνουμε επί τη βάση του περιεχομένου. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν και για ορισμένα άλλα θέματα όπως ε, τα διάφορα κινητά προϊόντα εκτός οδικού δικτύου. Δεν βρήκαμε λόγο για παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ε, βλέπουμε γιατί έχει κάνει τέτοια πρόταση η Κομισιόν. Γι' αυτό και δεν θα ζητήσουμε απόρριψη. Είναι κρίμα που κάνει μια δήλωση ο Κολγκέτη κάνει μια δήλωση και μετά χάνει την καλύτερη στιγμή που οι πράσινοι δεν το απορρίπτουν. Είμαι βέβαιο πω ο βοηθό θα του διαβιβάσει. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο, Πρόεδρε, γιατί ξέρω πω βιάζεστε και μπορώ να είμαι και γρήγορο εκτό από αυτή την ε, ε, μικρή το αστιάκι με τον συνάδελφο Κράμερ. Κύριε Ταταρέλα, εκτιμούμε αυτό που κάνετε, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι δεν προχωρά σωστά η Κομισιόν. Δεν λέμε μεν απόρριψη, αλλά δεν βλέπουμε το λόγο για αναβολή των θεμάτων. Δεν είμαστε υπέρ αυτών των τροπολογιών και απλώς ακολουθούμε την πρόταση της Κομισιόν. Και δεν ζητάμε αναβολή, ε, απόρριψη. Φαντάζομαι θα χαρείτε κάποιοι. Όλο. Πάντα μαθαίνουμε. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο για το θέμα αυτό. Ο κύριος Ρέντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει λοιπόν το λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας σε σχέση με την εργασία που έκανε ο κύριος Σταταρέλα εισηγητής σας, αλλά και σε σχέση με την πρόταση που κάνει, που πιστεύουμε ότι έχει νόημα. Πριν να η τελική απόφαση, που και που χρειάζεται αναθεώρηση της ισχύου σας κατάστασης. Και αυτό με φέρνει και στην παρέμβαση του κ. Κράμερα. Όταν υιοθετήθηκε η οδηγία το 2000, υπήρχαν ήδη κάποια ερωτηματικά σε σχέση με το κατά πόσο οι προδιαγραφές για τις εκπομπές των εξατμίσεων ήταν κατάλληλες για τα μικρά τρακτέρ. Γι' αυτό και συμφωνούμε ότι μπορεί να γίνει και περαιτέρω αναθεώρηση αν αυτό είναι απαραίτητο. Πάντως η εν γέννη είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά και υποστήριξη για την πρότασή μας. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κύριε Ρέντες. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 16 Ιουνίου. Στις 12. Αυτή την εβδομάδα. Όποιος θέλει να καταθέσει τροπολογίες για την έκθεση στα Ταρέλα μέχρι τις 16 Ιουνίου, ώρα 12 το μεσημέρι. Περνάμε λοιπόν στο 6 της μερίσιας διάταξης, το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και τον εξυγχρονισμό των ε, δημόσιων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η συγκεντριά μας είναι η ε, Όζα Βέστλοντ. Έχετε το λόγο για να κάνετε εισαγωγή στο θέμα αυτό. Ja, jag ska försöka, herr ordförande. Eh, Offentlig upphandling är ju ett brett område och jag tror att implementeringen trots ναι, πρόκειται για ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και νομίζω πως ε, η εφαρμογή γίνεται με, διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο ε, μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίε. Ε, κατά την άποψή μου, με βάση την εμπειρία μου, είναι ότι, ε, θα σας πω ότι συχνά η νομοθεσία αποτελεί εμπόδιο ε, για τις κρατικές προμήθειες. Υπάρχει δηλαδή καλή βούληση, αλλά δεν ε, είναι πολλά πράγματα δυνατόν να γίνουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Να επιβληθούν περιβαλλοντικά κριτήρια, ε, διατρέχει κανείς τον κίνδυνο να ε, διωχθεί ποινικά και κατά κάποιο τρόπο είναι ευκολότερο για τις τοπικές αρχές να μην χρησιμοποιήσουν αυτά τα κριτήρια και αυτό είναι κρίμα γιατί χρειάζεται να έχουμε βιώσιμα κριτήρια αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας στην Ένωση. Άρα λοιπόν συνέταξα αυτή τη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και νομίζω πως ε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στην αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να θαρρύνουμε ε, όσους ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις να κάνουν περισσότερο για το περιβάλλον. Κάτι που θα πρέπει εδώ να μας απασχολήσει είναι ότι η Κομισιόν περιμένει να δούμε εμείς ποιες είναι οι βασικές γραμμές, βασικά κριτήρια για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Εγώ έχω κρατήσει μια σχετικά ένα σχετικά χαμηλό προφίλ και με τις επαφές που είχαμε συναδέλφους φαίνεται πως όλοι συμφωνούν πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές ε, προδιαγραφές αλλά ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο γενικότερη κατεύθυνση για το πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτά και ίσως ε, ε, έτσι να θέσουμε περιβαλλοντικά κριτήρια και περιβαλλοντικά χαμηλά έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένα και να εμποδίσουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο στενά το κόστος του κύκλου ζωής και το κριτήριο της ε, καλύτερης τιμής ε, επίσης. Δεν νομίζω πως πάντοτε η χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να είναι το κριτήριο που θα χρησιμοποιείται, γιατί αυτό μας ε, εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε άλλα σοβαρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Μπορούμε να θέσουμε τεχνικές, τεχνικές προδιαγραφές, αλλά καλύτερα να πούμε ότι το περιβαλλοντικό κριτήριο είναι αυτό που θα επικρατεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επίσης το γεγονός ότι ε, αυτή τη στιγμή οι σχετικές διατάξεις ε, για τις κρατικές προμήθειες περιλαμβάνονται τα αυτό που μπορούμε να πάρουμε και να, ή να παραγγείλουμε για να έχουμε. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικέ επιπτώσεις και αντίκτυπο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σύνολο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος μιας υπηρεσίας. Ελπίζω πως η Επιτροπή θα με στηρίξει σε αυτό. Και τέλος, νομίζω πως μπορούμε να θεωρήσουμε διάφορα πράγματα αντιφατικά εδώ. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αντιφατικό είναι το τοπικά παραγόμενο, τοπικά παραγόμενο τρόφιμα. Πολλοί θέλουν να έχουν τρόφιμα τοπικά παραγόμενα για τα σχολεία, για τους ηλικιωμένους κτλ. Όμως σύμφωνα με τις αποφάσεις του 10 αυτό είναι αντίθετο με τις συνθήκες. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η νομοθεσία εδώ στην οδηγία, ωστόσο θα πρέπει κανείς να μπορεί να θεσπίσει κάποια κριτήρια όπως ε, ο αντίκτυπο στο κλίμα τη μεταφορά των τροφίμων, δηλαδή, μεταφορά, δηλαδή το αποτύπωμα μεταφοράς ε, των τροφίμων και δεδομένη τη κατάστασης πραγματικά είναι γελίο να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να μην επιβάλλουμε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό κριτήριο για το τρόφιμα, καθώς αυτό επηρεάζει το κόστος του κύκλου ζωής. Είναι μεγάλο το αποτύπωμα στο κλίμα και δεν είναι εύκολο να δει κανείς τι μεταφορές και τις εκπομπές. Προφανώς ένα κοτόπουλο που παράγεται 10-20 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που, που καταναλώνεται θα έχει λιγότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον από τα κοτόπουλα που φτάνουν από την Ταϊλάνδη. Θα πρέπει να είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξουν τέτοιου είδους απαιτήσει για περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και έπειτα δει κανείς ε, τις ντομάτες που παράγονται σε θερμοκήπια ή αυτούς που παράγονται ε, υπαίθριοι στην Ισπανία. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τα πράγματα και να λάβουμε υπόψη τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα που οφείλονται στη μεταφορά τροφίμων, τότε σίγουρα Εκείνοι που κάνουν τις ε, δημόσιες συμβάσεις σε τοπικό επίπεδο μπορούν να παίξουν ρόλο ε, στις κλιματικές αλλαγές. Αυτό δεν είναι δυνατόν ωστόσο σήμερα, είναι μια κατάσταση γελία που βασικά είμαστε υποχρεωμένοι να απορρίψουμε, μάλλον να αποδώσουμε μια σύμβαση σε κάποιον φορέα ο οποίος παράγει περισσότερες ε, εκπομπές. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Äh, Σας ευχαριστώ. Οι δημόσιες συμβάσεις νομίζω ότι αποτελούν 18% του ΑΕΠ. Μεγάλος όγκος ε, προμηθειών και συμβάσεων. Θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για τον ιδιωτικό κλάδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουμε διάφορους σκιώδες εισηγητές. Ο Γιάννος Όντα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα διότι στο πρώτο σημείο ήταν, είχε αντιστραφεί, ήταν αντιστραμμένη η κατάσταση. Δηλαδή εγώ ήμουν ο εισηγητής και εσείς ε, κυρία Βέσλουν και η Σκεώδης, η συγκήτρια, τώρα είναι το αντίστροφο ακριβώς. Λοιπόν, λίγοι μεταξύ των συναδέλφων θα γνωρίζουν ότι στα πλαίσια της πράσινης βίβλου η Κομισιόν έστειλε 114 ερωτήσεις προς τους ενδιαφερόμενους. Και μετά υπάρχει και μια άλλη πλευρά η οποία ε, καλύπτεται απόλυτα από την εισηγήτρια γιατί χρειάζονται αυτά τα μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις. Πολλοί λένε εγκρίναμε τη στρατηγική του 2020 με την Πρόκειται λοιπόν ε, για ε, ένα μέσο πολύ σημαντικό, εξυγχρονισμός δηλαδή των δημοσίων συμβάσεων για την Ευρώπη 2020, προστασία του περιβάλλοντος, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αλλαγή του κλίματος. Μπορούμε λοιπόν εμείς ε, να προσεγγίσουμε τους στόχους και μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις. Είμαι υπέρ της νομοδότησης της κυρίας Βέστλουγκ, Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στα σημεία 6 και 7. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μιλάμε για τον κύκλο ζωής και είναι πολύ σημαντικό να κερδίζει τη δημοπρασία, δηλαδή την, την ε, δημόσια σύμβαση, η προσφορά εκείνη που θα είναι πιο οικολογική. Δεν θα πρέπει να εκτιμάμε δηλαδή μόνο την χαμηλότερη προσφορά, αλλά και τις οικολογικές πλευρές. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε νέες σκέψεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Άλλο τώρα σε ένα νέο κανονισμό, σε μια νέα οδηγία πρέπει να λέμε σαφέστατα τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους εθνικούς νομοθέτες. Πρέπει να δίνουμε σαφείς ενδείξεις. Αν αφήσουμε όμως πολύ περιθώριο στα εθνικά κράτη, ορισμένα κοινοβούλια μπορεί να υλοποιήσουν το μέτρο πλήρω, άρα μερικώ ή άλλα καθόλου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ενιαίο εφαρμοστικό πλαίσιο. Χρειάζεται επίσης ομοιογένεια για όλα αυτά τα κριτήρια, τα νέα κριτήρια για τις δημόσιες συμβάσεις ούτως ώστε να τα στείλουμε εγκαίρως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όταν το πράσινο στοιχείο της δημοπρασίας είναι αυτό το οποίο βοήθησε στο να κερδιθεί η αγορά, τότε πρέπει να γίνεται έλεγχος ούτως ώστε ο, ο νικητής της δημοπρασίας αυτός που πήρε τη δημόσια σύμβαση να ελέγχεται ότι κρατάει τις υποσχέσεις του. Σύμφωνο με αυτά που μας είπε λοιπόν η κυρία Βέστρουγκ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βέστρουγκ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε στο σχέδιο αυτό που περιλαμβάνει πολλά σημαντικά στοιχεία με τα οποία συμφωνώ. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της ε, στρατηγικής για το 2020, είναι σημαντική, σημαντικό μέσο οι δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να πετύχουμε περιβαλλοντικώς ε, φιλικά ε, προϊόντα και υπηρεσίες. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν υπόψη περιβαλλοντικέ διατάξει υπόψη κατά την ανάθεση συμβάσεων. Έχω όμω κάποιε προτάσει να κάνω. Καταρχά, η διατύπωση στο σημείο 4 δεν είναι σαφή. Δεν καταλαβαίνουμε κατά πόσον θα πρέπει να αποτελεί αυτό τμήμα των κριτηρίων ή όπως προβλέπει η οπω προβλεπει νομοθεσία ε, θέμα τεχνικής τεχνικης προδιαγραφη σω θα μπορούσε να μα βοηθήσει και να το διευκρινίσει αυτό η συγγήτρια, γιατί θεωρώ ότι αν συμπεριληφθεί στα κριτήρια θα μπορεί να προωθηθεί η κοινοτομία. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν, λέτε, οι διατάξεις αυτές σε, όλα, σε όλες τα συμβάσεις. Αυτό δεν συνάδει λίγο με το 7, γιατί μπορεί να υπάρχουν συμβάσεις που δεν είναι περιβαλλοντικώς σχετικές. Άρα αυτό θα πρέπει να λεφθεί υπόψη όχι σε όλες τις συμβάσεις, μόνο στις σχετικές συμβάσεις. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει η λύση του να λεφθεί υπόψη αυτό στο, στις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, το κόστος κύκλου ζωής θα πρέπει και αυτό να λεφθεί υπόψη όπως αναφέρει στο σημείο 6 η συγγήτρια, αυτό θα ήταν ε, μια δυνατότητα, όχι υποχρέωση. Θα πρέπει να συζητήσουμε, θεωρώ, τη δυνατότητα να καταστεί υποχρεωτικό. Γιατί θα είναι λογικό αυτό, γιατί μπορεί ένα προϊόν να είναι πιο ακριβό από ό,τι φαίνεται εκ πρώτη όψεως, αν συμπεριληφθεί και το κόστος ε, απόρριψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μία μέθοδο για τον υπολογισμό του κόστους αυτού και να βοηθήσει έτσι τις αρχές να επιλέξουν τις καλύτερες λύσεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση μεταξύ δημοσίων συμβάσεων και των περιβαλλοντικών στόχων. Να μην ξεχνάμε όμως και το θέμα του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία στο σημείο αυτό προκειμένου να μην βλάψουμε τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις μας δεν θα δυσκολέψουν την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τέτοιες ε, δημόσιες ε, συμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος. Thank you, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το θέμα, για, όπως είπατε νωρίτερα. Και η ε, ενημέρωση αυτών των κανόνων μας δίνουν μια ευκαιρία να υποστηρίξουμε την ισορροπία μεταξύ βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος στην Ένωση. Όπω υπόθηκε, ήδη είχαμε μια συνάντηση και διαπιστώσαμε μεγάλο βαθμό συμφωνία. Εγώ καλωσορίζω τη γνώμη τη εισηγήτρια και συμφωνώ με το μεγαλύτερο τμήμα. Αντίθετα με τον προηγούμενο μιλητή, συμφωνώ απόλυτα ότι οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλε τι συμβάσει δημοσίων προμηθειών προμηθειών, κρατικών Βέβαια, Μπορεί να έχουμε καλές προθέσεις, αλλά να μην είναι εύκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά και τελικά να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα αποθαρρύνοντας τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις ποσοστώσεις. Συμφωνώ ότι το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα πρέπει να επιλέγεται μόνο αν αιτιολογείται ε, και με βάση τις τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και απαιτήσει. Ε, τότε και μόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το θέμα της τιμής. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει διεύρυνση της συνένεσης και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο, όπως είπε η συγκήτρια, εξασφάλισης ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα ευνοούν τις τοπικές επιχειρήσεις, γιατί αυτό έχει μόνο ωφελεί την τοπική οικονομία και θέσεις απασχόλησης, αλλά και καταπολεμεί τις κλιματικές αλλαγές και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα, καθώς και έχει θετικές επιπτώσεις στους τομείς αυτής. Στη δική μου περιφέρεια, στην Ουαλία, περίπου το ίμιση των υπηρεσιών που αγοράζονται από το δημόσιο τομέα αγοράζονται από προμηθευτές που έχουν έδρα στις, στην Ουαλία. Ελπίζω πως αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, αλλά είναι κάπως προβληματικό γιατί στο άρθρο 101 της λόγω του άρθρου 101 της συνθήκης όλοι συμφωνούμε με την να ευνοούμε τους τοπικούς εργαζόμενους, να αγοράζουμε τοπικά τρόφιμα, να πηγαίνουμε στα τοπικά σχολεία κτλ. Και θα προσπαθήσω με την εισηγήτρια να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε το θέμα μέσω τροπολογιών ώστε κάτι τέτοιο να γίνει στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Evans για να κουδάκεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Νομίζω πως ε, ακολουθεί η σωστή γραμμή στο... θα στηρίξουμε το μεγαλύτερο τμήμα της εκθεσής της. Έχουμε κάνει κάποιες τροπολογίες. Βασικά όσον αφορά την θέση ότι τα συμφέροντα των κρατών μελών θα πρέπει να συνδυάζονται με το καλό της Ένωσης και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να τα συνδυάσουμε αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς. Συμφωνώ επίσης με τους φιλελεύθερους ε, συνάδελφους ότι βασικά πρόκειται για οδηγία που αφορά την ιστορική αγορά και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη να κρίσουμε το περιβάλλον γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργήσουν όλα αυτά πολύ καλά. Εμείς εργαζόμαστε με σεβασμό των θέσεων των κρατών μελών όσον αφορά το πρωτογεν... το... τα συμφέροντά τους. Έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικοί προβληματισμοί στην παράγραφο 7. Όμως δεν είναι ότι μόνη μας ανησυχία, θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην προσέγγισή μας. Επίσης πιστεύουμε ότι η πολιτική θα πρέπει να μπορεί να ε, έχει και κινητούς στόχους, ενώ αν έχουμε υποχρεωτικούς στόχους, κάτι τέτοιο θα περιόριζε το πώς θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία ενθάρρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, να συμμετέχουν σε αυτές τις ε, συμβάσεις ε, με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Εν γέννη λοιπόν να υποστηρίζουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Η Σαμπίν Βίλτς. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά της. 16% του ΑΕΠ της Ένωσης είναι οι δημοπρασίες. Δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει τεράστια δυνατότητα λοιπόν να επηρεάσει και ε, συμπεριφορές, οικονομικές συμπεριφορές ή περιβαλλοντικές συμπεριφορές. Κοιτώντα την πράσινη βίβλο που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπω ότι υπάρχουν ε, βασικά προβλήματα. Υποστηρίζω λοιπόν την πρασινη βιβλο που εχει καταθεσει η ευρωπαικη επιτροπη βλεπω οτι υπαρχουν βασικα προβληματα υποστηριζω λοιπον την εισηγητρια με το καλό σχέδιο γνωμοδότησης που μας παρουσίασε. Είναι πολύ σημαντικό για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις προσπάθειε για την προστασία του κλίματος στι δημόσιε συμβάσει να προσέχουμε προκειμένου να μην επιλέγουμε μόνο τον οικονομικά πιο ευνοϊκό υποψήφιο. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όλος ο κύκλος ζωής ε, του προϊόντος και οι επιπτώσεις ε, στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το ανέφερε αυτό η κυρία Βέστλουντ. Όπως σωστά αναφέρει η κυρία Βέστλουντ, ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προβάλλει τα πλέον εκτήματα συμπεριλήψης, ε, περιβαλλοντικών ε, παραγόντων. Και κυρίως είναι μακροπρόθεσμα αυτά τα ωφέλη, γιατί συχνά δυσκολευόμαστε ως πολιτικοί να ε, αφήσουμε κατά μέρος το βραχυπρόθεσμο προς όφελος του μακροπρόθεσμου. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι εργασιακές συνθήκες, γιατί η πίεση στις τιμές προκαλεί σε πολλές επιχειρήσεις ε, κάθε διπτώση των εργασιακών συνθήκων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει την εξουσία της προκειμένου οι μισθοί να τηρούνται τα μισθολογικά μάλλον όρια και οι εργασιακοί όροι οι κοινωνικοί όροι. Νομίζω λοιπόν ότι θα καταθέσουμε μια καλή ε, γνωμοδότηση και να δούμε τι θα απομείνει όταν θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους και οι υπόλοιπε επιτροπές που συμμετέχουν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο ακόμα ομιλητές. Σοφή Οκουνή. Euh, Σύντομα πολλά πράγματα υπόθηκαν. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω για όλη αυτή τη δουλειά. Οι, δημοπρα... οι δημόσιες συμβάσεις είναι το 16% όλου του ΕΠ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προβληματική. Και υπάρχει ένα σημείο που το θεωρώ ουσιαστικό, έστω και αν πρόκειται για οδηγία εσωτερικής αγοράς και όχι απόλυτα συμβατή, δηλαδή με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μία από τις μεγάλες δημοπρασίες που έγιναν στην Πολωνία πρόσφατα, μία από τις δημόσιες συμβάσεις δηλαδή, την κέρδισε μία κινέζικη επιχείρηση για την κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου με κοινοτικά κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτές τις προβληματικές, διότι οι Κινέζοι σήμερα μπορούν να ε, κατακτούν τις αγορές μέσα από τις ε, δημο, δημοπρασίες χωρίς όμως δικές μας επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κινέζικες δημόσιες συμβάσεις. Και δεν ξέρω κατά πόσο οι Κινέζοι μπορούν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες μας από περιβαλλοντική Κυρία Γιούζο, όχι, α, Κυρία Βέσλουγκ, θέλει να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει καταφτάσει ο Επίτροπος Ντάλι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους συναδέλφους και τα σχόλιά τους. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλή γνωμοδότηση. Όλοι οι συνάδελφοι συνέβαλαν στην παράγραφο 4 στα Σουηδικά. Είναι σαφές ότι αναφέρεται ότι οι περιβαλλοντικές ε, ανησυχίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλες ε, τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Και στην παράγραφο 4 γίνεται μια απόπειρα να πούμε ότι είτε θα πρέπει να υπάρχουν περιβαλλοντικές ε, διατάξεις στις τεχνικές προδιαγραφές ή να χρησιμοποιηθούν περιβαλλοντικές πτυχές σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ανάθεσης. Ίσως σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτό θέλω να εκφράσω στο σημείο αυτό. Ίσως θα μπορούσα να αλλάξω τη διατύπωση κάπως. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Άζα Βέστλουντ. Το θέμα αυτό του εξυγχρονισμού των δημοσίων συμβάσεων από τις ε, Θεωρούμε από πλευρά στην Επιτροπή, Επιτροπής μας ότι χρειάζεται πιο πολύ βιωσιμότητα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 16 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι 16 Ιουνίου, όποιος θέλει να καταθέσει τροπολογίες. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Confidustria από την Ιταλία. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, Συνεδριάσατε ετησίως εδώ στις Βρυξέλλες και βλέπω ότι παρακολουθείτε λοιπόν ένα μικρό τμήμα της Επιτροπής μας. Και το επόμενο θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε ορίζω τον Επίτροπο Τζον Ντάλι, Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ένα θέμα το οποίο μας άγγιξε ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ο ιός Έχεκ, ο οποίος ε, έπληξε τη Γερμανία αλλά και πολλές άλλες ε, χώρες και προκάλεσε μεγάλη ζημιά και στη Γεωργία προκάλεσε μεγάλες αναταραχές. Στο Στρασβούργο είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε διεξοδικά. Ήταν ενδιαφέρον που ακούσαμε ότι σήμερα θα γινόταν η σχετική παρουσίαση. Πρόκειται για ένα θέμα, ένα καινούργιο θέμα Πέρσι είχαμε την ε, γρήπη των χείρων, τον ΙΤΑ 1 που κινητοποίησε την Ευρώπη. Φέτος είναι η σειρά του ΕΧΕΚ, το βακτήριο του ΕΧΕΚ. Και βλέπουμε πόσο μικρή σημασία έχουν τα σύνορα βλέπουμε πως πλήττονται οι διάφοροι οικονομικοί τομείς, πόσο μεγάλη ζημιά μπορούν να υποστούν, αν δεν υπάρχει η βέλτιστη διαχείριση. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο πολλοί ε, συνάδελφοι ανέφεραν ένα χάος στην επικοινωνία. Στην περίπτωση της Γερμανίας έχουμε ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης όπου 16 κρατήδια, ομοσπονδιακά κρατήρια, κρατήδια έχουν ε, και τα Υπουργεία Υγεία τα εργαστήριά τους. Έχουμε το εθνικό επίπεδο, το ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να αντιδρούμε το σύντομότερα δυνατόν, να διευκρινίζουμε τέτοιες ε, καταστάσεις προς όφελος και του κόσμου ασφαλώς, αλλά και προς όφελο του εμπλεκόμενου κλάδου, προς όφελος της οικονομίας. Επίτροπε, σα δίνω το λόγο για να μας αναφέρετε πώς βλέπει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια <coughs> μαθήματα θα πρέπει να εξάγουμε. Έχουμε φυσικά και την υπηρεσία στην Στοκχόλμη για το κέντρο, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ε, πρόληψη των νόσων. Τι θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν για να μην μας παίρνει τρεις-τέσσερις εβδομάδες μέχρι να υπάρχει κάποια βεβαιότητα για τα αίτια και για να μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα προς τους πολίτες μας. Έχετε το λόγο. Well, thank you very much, uh, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε για ενημέρωση όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις μετά από την, ε, το ξέσπασμα της επιδημίας, η κόλλη και μετά από τις δηλώσεις μας στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Όλοι μας ανησυχούμε ιδιαίτερα για το βαρύ φορτίο ε, θανάτων ε, και ασθενών που προκάλεσε αυτή η τροφική επιθυμία και πρέπει ακόμη μια φορά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όσους έχασαν δικούς τους. Υπάρχουν τώρα 3.000 ε, ε, περίπου περιστατικά 120 άνθρωποι δεν έχουν άσχημες εξελίξεις και επιπλοκές το ε, σε αυτή την επιδημία οφείλονται 25 θάνατοι μέχρι στιγμή στην Γερμανία και ένα στην Σουηδία. Δυστυχώ μπορεί να υπάρξουν και άλλοι θάνατοι αυτέ τι μέρε λόγω τη μακρά περίοδου επόαση του Τη ασθένειας και γιατί μπορεί η αγωγή που δίνεται να μην μπόρεσε να σώσει αυτούς που έχουν μολυνθεί. Βόρεια του Αμβούργου είναι το επίκεντρο και πολλές από τα, πολλά από τα περιστατικά αφορούν είτε Γερμανούς υπηκόους που ταξιδεύουν είτε ανθρώπους που επισκέφθηκαν τη Γερμανία ε, στην περιοχή αυτή. Τώρα στραφώ στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτή την επιδημία. Καταρχήν δραστηριοποιήσαμε άμεσα όλα μας τα δίκτυα που είναι υπεύθυνα για την αρμόδια για την διαχείριση κρίσεων όταν λάβαμε την πρώτη κοινοποίηση από τη Γερμανία στις 22 Μαΐου. Το δίκτυά μας ήταν σε καθημερινή επαφή και μας επέτρεψαν την έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Καθημερινές δε επαφές έχουμε με τις αρχές δημόσιας υγείας και τη ασφάλεια των τροφίμων στα κρατημέλη για να συζητάμε την εξέλιξη της επιδημίας. Τα μέτρα υγείας που ελήφθησαν για την πρόληψη της μόλυνσης και την αγωγή των ασθενών τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ε, για τα τρόφιμα και τις οτροφές ε, μας έχουν δώσει στέρεα βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών. Εμεί ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη Ασθενειών για τον Έλεγχο να προβεί σε επιστημονική εκτίμηση που ενημερώνεται καθώ εξελίσσεται η κατάσταση. Το κέντρο αυτό επίση είχε αναπτύξει σε, στο επίπεδο της, ε, του, οργανισμού για την, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Τροφίμων συμβου, ε, συμβουλέ που δίνονται στο, δημόσιο, στο κοινό συγγνώμη, και υπάρχουν διθέσιμε σε όλε τι γλώσσε της Ένωσης. Έχουμε καλέσει επίσης το αρμόδιο αυτό οργανισμό να φτιάξει έναν κατάλογο καλύτερο πρακτικών. Η Κομισιόν ζήτησε από την, αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων να δώσει συμβουλές για διάφορα, περι διάφορες θέματα συμπεριλαμβανομένου του επίπεδου μόλυνσης ε, των νοπών λαχανικών. Ήδη σε μέσα σε δύο μέρες ε, προέβησαν σε αυτές τις συστάσεις. Πρώτον ε, είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής υγιεινής σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Επίση έχουν γίνει έρευνες εκεί που είχε εντοπιστεί σε παλιότερα χρόνια το συγκεκριμένο ε, βακτηρίδιο. Τέλος, η βοήθεια των εμπειρογνωμόνων της ε, ΕΦΣΑ, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στα Τρόφιμα, ήταν κρίσιμη όσον αφορά τη... τον εντοπισμό των φύτρων που βρίσκονταν στην πηγή της ε, επιδημίας. Σε χρόνο ρεκόρ δε αναπτύχθηκε μέθοδος για τον εντοπισμό του βακτηριδίου E. coli από τις 60 ε, μέρες στις 48 ώρες περιορίστηκε ο χρόνος εντοπισμού του βακτηριδίου. Οι ενημερώσεις δε της Κομισιόν μαζί με το συγκεκριμένο δίκτυο ενημέρωσης αλλά και τις αρχές ασφάλειας των τροφίμων είναι διαρκείς και φυσικά ενημερώνουμε το site μας για τις εξελίξεις αυτής της επιδημίας. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές να επιστηρίξουν αυτή την επιστημονική ανακοίνωση ώστε να περιοριστεί ο άσκοπος φόβος. Ε, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η Κομισιόν μαζί με τους διάφορους οργανισμούς της εξακολουθεί να δουλεύει σκληρά με, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ε, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την επιδημία. Την ε, Κυριακή 5 Ιουνίου, ειδικοί επιδημιολόγοι για τις Ασθένειε ε, που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων πήγαν στην Γερμανία για να βοηθήσουν ε, με τις συνεχιζόμενες έρευνες για τον εντοπισμό της πηγής. Ε, Στι 6 Ιουνίου η κατάσταση συζητήθηκε με τους υπουργούς στο, Υπουργείο, στο Συμβούλιο Υγείας. Ζήτησε από τη Γερμανία να, να ενισχύσει τους ελέγχους για να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας. Και επίσης ε, και να εντοπιστούν τα αίτια. Την Τρίτη, στις 7 Ιουνίου, συζητήσαμε στην Ολομέλεια για το θέμα της επιδημίας αυτής, όπου τονίστηκε ότι κάθε προσπάθεια θα πρέπει να γίνει για τον εντοπισμό της πηγής της ρήπασης, της μόλυνσης. Επίσης, κατέστησα σαφές ότι τα μηνύματα προς το ευρύ κοινό είτε προέρχονται από ειδικού είτε από πολιτικού, θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία για να μην επικρατεί πανικός. Ε, την ίδια μέρα ο Επίτροπος Τσιόλος και εγώ ε, μιλήσαμε στο Συμβούλιο Γεωργίας στο Λουξεμβούργο που διοργάνωσε η Ουγγρική Προεδρία για να συζητηθεί το, η επιδημία η κόλλη και οι οικονομικές της ε, επιπτώσεις. Στις 8 Ιουνίου παρακολούθησα το σύσκεψη των Υπουργών Γεωργίας όλων των κρατηδίων καθώς και επισκέφθηκα το Βερολίνο και το την ομάδα κρίσης. Τους παρότριναν να κάνουν μόνο ανακοινώσεις με βάση επιστημονικά ασφαλή στοιχεία. Επί τη βάση λοιπόν επιδημιολογικών στοιχείων στις 9 Ιουνίου οι γερμανικές αρχές μπόρεσαν να εντοπίσουν ένα αγρόκτημα που παράγει διάφορα φύτρα φασολιών ε, και όπου από ό,τι φαίνεται ήταν η πηγή του επιδημίας. Στις 11 του μηνός οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν τα απορίσματα μέσω εργαστηριακών ελέγχων. Η συγκεκριμένη σειρά ε, η βακτηριδίου η κόλλη που είναι υπεύθυνη για την μόλυνση των ανθρώπων ε, εντοπίστηκε σε, αυτήν, σε αυτό το αγρόκτημα παραγωγής φύτρων. Ελπίζω πως, ε, τα, πως οι κύριοι βουλευτές συμφωνήσουν ότι είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η εξέλιξη. Έχει εντοπιστεί η πηγή και επιδημιολογικές, ε, τα επιδημιολογικά πορίσματα υποστηρίζονται από εργαστηριακούς ελέγχους. Φυσικά θα συνεχίσουμε την έρευνά μας ώστε να ολυρώσουμε την εικόνα της σύνδεσης ανάμεσα στους ανθρώπους που αρρώστησαν, τα ε, το συγκεκριμένο αγρόκτημα αλλά και ε, διάφορα ε, και πώς μάλλον προχώρησε η σειρά αυτή του βακτηριδίου μέσα στην τροφική αλυσίδα. Όπως σας έχω ήδη δηλώσει, η Κομισιόν με τα κρατημέλη θα αποκομίσουν διδάγματα από αυτή την κρίση για το πώς θα βελτιωθεί περαιτέρω. Η χρήση του συστήματος έγκυρης προειδοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές να μην προτρέχουν, να μην διαδίδουν ε, νέα πριν αυτά να έχουν ε, επικυρωθεί και ελεγχθεί. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα για τους παραγωγούς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Αυτή η επιδημία αποδεικνύει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να διερευνούν ε, με δελεχώς τις, πιθανούς, τις πιθανές πηγές μόλυνσης και να προβαίνουν έπειτα στην έγκαιρη προειδοποίηση. Ωστόσο, όπως έχω ήδη δηλώσει στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι σε όλες μας τις αντιδράσεις δεν θα προκαλούμε φόβο Στου ηθήνοντε για τη λήψη αποφάσεων, ώστε αυτοί να μην λάβουν, να μην λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις που θα έπρεπε να παίρνουν για να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών τους. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, τότε μπορούμε να μάθουμε από τα διδάγματα αυτή τη κρίσης και να βελτιώσουμε περαιτέρω τη λειτουργία των συστημάτων μας. Συντονισμούς, σαφείς γραμμές ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτελούν τον πυρήνα Τη δυνατότητά μα να είμαστε αποτελεσματικοί σε τέτοιε περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε πολλά σε αυτό το επίπεδο και επίση να σα αναφέρω την ανησυχία μου σε σχέση με τι ισχύουσε απαγορεύσει για ορισμένα προϊόντα. Θέλω να τονίσω άλλη μια φορά ότι το ξέσπασμα τη επιθυμία περιορίζεται γεωγραφικά σε μια περιοχή που ε, περικλεί την πόλη του, του Αμβούργου. Δεν υπάρχει λόγο λοιπόν να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό το φως του εντοπισμού της ε, πηγής νομίζουμε πως η υπαγόρευση οποιοδήποτε προϊόντος είναι δυσανάλογη, άκερη. Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν δουλέψει σκληρά για να εφαρμόσουν την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στις 10 Ιουνίου Παρασκευή ανάμεσα στον Πρόεδρο Παρόζο και τον Ρώσο Πρόεδρο Δημήτρη Μετβέντεφ στην διάσκεψη κορυφής ΕΕ Ρωσίας στο που προβλέπει άρση της απαγόρευσης εισαγωγής ευρωπαϊκών λαχανικών, νοπών λαχανικών και την εισαγωγή εγγύσεων. Από τη στιγμή που πετεύχθη η συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν και οι Υπηρεσίε της προώθησαν συγκεκριμένη πρόταση προς τις ρωσικέ αρμόδιες αρχές. Σήμερα δεν έχουν κοινοποιήσει ότι εν ώψη της Μάλλον ότι αυτή η ε, παρότρινση μπήκε στην συμφωνία Μπαρόζο Μετβέντεφ. Δεδομένου των σημαντικών ε, πορισμάτων και της ανέβρεσης το πηγής της επιδημίας ε, και του περιορισμού αυτής στις φύτρες θεωρούμε ότι εμπίπτει η πρότασή μας στη συμφωνία μεταξύ Μπαρόζο και Μετβέντεφ, Πλούσουμε να επανεξετάσουν οι ρωσικές αρχές αυτή την πρόταση ώστε η εξαγωγή των όπών προϊόντων να επαναληφθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Τέλο, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά την οικονομικό αντίκτυπο που έχει αυτή η κρίση στου γεωργού και κυρίω στου παραγωγού λαχανικών. Και γι' αυτό συνεργάζομαι στενά με τον συνάδελφο Τσόλο για να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε των παραγωγών που επίση επλήγησαν από την επιδημία. Η Κομισιόν ε, συνεργάζεται στενά με τα κρατη με ε, κοινό στόχο να λήξει αυτή η επιδημία όσο γίνεται πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Yeah, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντάλη, για την παρουσίαση αυτή, για την τρέχουσα κατάσταση σήμερα, 3η 14 Ιουνίου. Ήσασταν πάρα πολύ απασχολημένος στις τελευταίες εβδομάδες, όπως βλέπουμε και από τις σημειώσεις σας ε, ε, απανοτές συνεδριάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ακολουθήσει η συζήτηση τώρα με τους βουλευτές της Επιτροπής μας. Και τώρα να το γυρίσω στα γερμανικά, λέει ο Πρόεδρος. Είπατε να μην ε, βιαζόμαστε και να μην... Ε, σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση προς το κοινό. Αυτό φυσικά ίσως να είναι ευσεβής πόθος, γιατί αυτό είναι και θέμα αρμοδιότητας, το ποιος θα ε, ενημερώνει το κοινό. Υπάρχει άραγε σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμός με, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, την δημοσίευση ανακοινώσεων προς το κοινό. Δεν είμαστε ΙΠΑ, ΙΠΑ έχουν μία αρχή για την ε, καταπολέμηση των νόσων. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου, του ΕΚΠΕΝ. Και έτσι να αποδείξουμε στους πολίτες ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ Ευρώπη. Χτες αναφέρθηκε ότι ίσως οι σπόροι για τα φύτρα αυτά να αποτέλεσαν την πηγή της μόλυνσης και δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση των σπόρων αυτών. Ήταν από το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ασία, από την Αφρική. Εδώ τίθεται και το θέμα της ανιχνεσιμότητας, όπως και το θέμα της ανιχνεσιμότητας των τροφίμων. Αυτό αφορά και θέματα πληροφόρησης για τα τρόφιμα και αυτό αποτελεί αντικείμενο τρομερούς διαλόγου. Οι Υπουργοί Γεωργίας θα ασχοληθούν με θέματα αποζημίωσης των γεωργών. Η αντίδραση της Ρωσίας καταδεικνύει πόσο ευαίσθητα είναι τα ζητήματα αυτά. Και όσο δυσανάλογη και αν φαίνεται η απόφαση που ελήφθησε να απαγορευτούν οι εισαγωγές από την Ευρώπη, θα πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι η Μόσχα ουσιαστικά σκοπό έχει την προστασία της υγείας των πολιτών της. Βλέπουμε λοιπόν ε, πώς αντιμετωπίζεται καθολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα των τροφίμων αποτελεί μια βόμβα η οποία μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει πολλές παράπλευρες ε, ζημιές. Η κυρία Πιλάρα Γιούζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Ε, εγώ είμαι σίγουρη ότι όλες οι υπηρεσίες της Κομισιόν εργάστηκαν πάρα πολύ και εσείς ε, μαζί με τους συναδέλφους σας αφιερώσατε πολλές ώρες γύρω από το θέμα. Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε με την έρευνα και να μάθουμε πώς το, το βακτηρίδιο ή κόλλη έφτασε μέχρι τους σπόρους ε, της σόγιας. Δεν πρόκειται για φυτολογικό παθογόνο. Ε, κάποια στιγμή έφτασε τις ε, φύτρες της όγιας μέσα από κάποια επεξεργασία. Πρέπει να μάθουμε πώς για να μπορέσουμε να λάβουμε και τα αντίστοιχα μέτρα. Λέτε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε και να μην, ε, για να μην δημιουργηθούν οικονομικά προβλήματα. Μα κοιτάστε, αυτό, ήδη το κακό έγινε. Η, κοινωνική πίεση ήταν τέτοια που την προηγούμενη εβδομάδα στο εστιατόριο Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο εστιατόριο δίπλα, δηλαδή στο, στο κτίριό μας του Στρασβούργου, υπήρχε μια πίσα που έλεγε ότι εδώ δεν έχουμε ισπανικά προϊόντα, ισπανικά τρόφιμα. Λοιπόν, μαθήματα πρέπει να, να ανασύρουμε, διδάγματα, να μάθουμε. Η αρχή της προόληψης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Δεν μπορούμε εμείς να, κάνουμε λάθος, να, δίνουμε λάθος και βιαστικές πληροφορίες μόνο στο όνομα της αρχής της πρόληψης. Θα πρέπει να δούμε τον 16 του 2011 κανονισμό για την ε, έγκαιρη επέμβαση. Πρέπει να ενημερώσουμε τους αρμόδιους ε, στην τροφιμική αλυσίδα και επίσης οι, τροφιμικές, ε, οι, συναγερμοί για τον κίνδυνο των τροφίμων δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικού πολέμου, πράγμα το οποίο έγινε. Και πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα αποζημίωσης και στο κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχουμε μόνο έναν συνομιλητή. Αυτό το οποίο συνέβη δεν πρέπει να ξαναγίνει πρόκειται για ένα δυσάρεστο επεισόδιο, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε όλα τα εκκρεμή προβλήματα και να τελειώνουμε με την έρευνα. Να μην ξεχνάνε οι γερμανικές αρχές και οι γερμανοί επιστήμονες να μην ξεχνάνε ότι πρέπει να βρεθεί η ρίζα αυτή της μόλυσης από αυτό το βακτηρίδιο, το E. coli είναι γνωστό εδώ και 15 χρόνια. Πρέπει λοιπόν εμείς να διαπιστώσουμε πώς έφτασε, πώς μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ευχαριστώ κυρία Γιούζο. Το να ψάχνει κανείς την αιτία είναι σαν να ψάχνει τελικά μια αμπελώνα στον αχυρώνα. οι πρώτες υποψίες ήταν λάθος. Ε, και έπληξαν τελικά τα ισπανικά αγγούρια, λάθος ήτανε. Καλόπιστο όμως. Το λάθος, αλλά λάθος ήτανε. Ο κύριος Λίζε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Ντάλη που είναι εδώ. Είχαμε μια ωραία συζήτηση μαζί του και την προηγούμενη εβδομάδα τον ευχαριστώ γιατί στην αρχή της τοποθέτησής σας κύριε Επίτροπε εκφράσατε αλληλεγγύη και τα συλληπιτήριά σας προς τα θύματα. Στην αρχή της ε, χρονιάς είχαμε το σκάνδαλο της διοξίνης Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και ένα σωρό θύματα, δεν είχαμε μόνο προμάρα. Κάτι πήγε στραβά, είπανε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αρχές του Αμβούργου πρώτα ενημέρωσαν ε, την κοινή γνώμη για τα ισπανικά αγγούρια και πολύ πιο αργά ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν μία συντονισμένη διαδικασία θα μπορούσε να μας είχε βοηθήσει να διαπιστώσουμε αμέσως την αιτία. Αλλά προσοχή. Δεν πρέπει εμείς να δίνουμε, θα πρέπει μάλλον να δίνουμε πληροφορίες στην κοινή γνώμη μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα. Βέβαια, ας φανταστούμε εμείς την αντίθετη περίπτωση ότι πάλι ύποπτα ήταν τα ισπανικά αγγούρια και δεν το είχαμε ανακοινώσει στην κοινή γνώμη. Ποιος πολιτικός θα αναλάμβανε την ευθύνη για όλους αυτούς τους ασθενείς στην εντατική παρακολούθηση και όλους τους θανάτους που επακολούθησαν. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να έχουμε ανοιχτά όλα αυτά τα κανάλια πληροφόρησης και μετά να διαπιστώνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την πραγματική αιτία. Αν υπάρχει υποψία για ένα εργαστήριο, ε, αν μάλλον συγγνώμη ένα εργαστήριο έχει την υποψία δεν πρέπει να περιμένει 100% να είναι σίγουρο για να το ανακοινώσει. Τα αντιβιωτικά εδώ είναι, δεν έχουν αποτέλεσμα. Ίσα ίσα επιβαρύνουν την κατάσταση. Και του χρόνου μπορεί να έχουμε μια άλλη περίπτωση, πάλι με ένα βακτηρίδιο που να αντέχει στα αντιβιωτικά και το οποίο να ανίατο. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο τον Μάιο ε, ε, ε, ψήφισε ένα ψήφισμα για την αντοχή στην, στα αντιβιωτικά. Ρωτώ την Κομισιόν, τι κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση Ευχαριστώ Πρόεδρε και σε ευχαριστώ Επίτροπε που μας δίνετε αυτήν την ενημέρωση μία μόλις εβδομάδα μετά από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Είπατε ότι πρέπει να μάθουμε διδάγματα από την για την επικοινωνία και ε, σημαντικό φυσικά γιατί όλοι εύκολα μπορούμε να αρχίσουμε να κριτικάρουμε και να λέμε πως δεν βρέθη αρκετά σύντομα η πηγή αυτού του βακτηρίου αλλά πραγματικά είναι σαν να ψάχνεις ψήλου τάχυρα. Συμφωνώ με τον Επίτροπο και είμαι βέβαιος ότι όλοι προσπαθούσαν να βρουν την πηγή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά εντωμεταξύ η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι δύσκολο να βρει κανεί την πηγή, αλλά ενώ ψάχνουμε όλη την πηγή είναι σημαντικό ε, να γίνει η επικοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί πανικός και ταυτόχρονα να μην αισιοποίησουμε κιόλα. Συμφωνώ με τον κύριο Λίζε ότι αν το αντιστρέψουμε και βρούμε το επιχείρημα και βρούμε καλά επιχειρήματα ότι η πηγή μπορεί να είναι για τα αγκούρια, όντω πρέπει να το πει ότι για την ώρα, ναι, καλύτερα να είμαστε ασφαλεί και μην τα τρώμε. Δεν συμφωνώ ότι ήταν πολύ σοφό να πούμε ότι βρέχονται από τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό δεν χρειαζόταν, ε. Μπορούσε κανείς να πεις ε, τα αγκούρια εν γέννη, χωρίς να πει από τα ποια αγκούρια ποιας εθνικότητα. Και φυσικά ένα παραπάνω αφού δεν ήταν βέβαιο. Η επικοινωνία λοιπόν είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι σημαντικό και για εσάς. Αλλά είπατε ότι πρέπει να μάθουμε, αλλά κάπως αόριστα το είπατε αυτό, δεν είπατε τι να μάθουμε. Αν δείτε πώς έγινε η επικοινωνία αυτή τη στιγμή στην Γερμανία, ήταν σαφώς ότι οι γραμμές ε, επικοινωνίας είναι πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους. Εντοπίστηκε σε ένα νοσοκομείο, πάει σε μια υπηρεσία τοπική για την υγεία, έπειτα στην περιφερειακή, έπειτα στην ομοσπονδιακή, που είναι το Ινστιτούτο Ρόμπερ Κόχ και μετά φτάνει στην Ένωση. Πολλά πολλά στάδια δηλαδή πριν να φτάσει στο επίπεδο το κοινοτικό, ότι έχουμε πρόβλημα. Και νομίζω εδώ η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει κάποιες προτάσεις ώστε να είναι πιο γρήγορη η επικοινωνία από ό,τι έγινε τώρα στη Γερμανία. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα κεντρικό οργανισμό καταγραφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι από τη στιγμή που εντοπίζετε το πρόβλημα θα, εντοπ... θα, δια... θα διαβιβάζετε αμέσως αυτόν τον οργανισμό γιατί φορτικά θα αργούμε, θα καθυστερούμε και αυτό είναι προβληματικό όταν έχουμε να κάνουμε επίγουσες ε, περιπτώσεις. Αν η Κομισιόν λέει λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε από την επικοινωνία ε, θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς μαθήματα, διδάγματα έχετε αποκομίσει ώστε να είναι πιο σύντομη η επικοινωνία και ότι θα υπάρξει κάποιο είδος κεντρικής καταγραφής ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ξέρουμε τι συμβαίνει και πότε όταν κάτι γίνεται σε νοσοκομιακό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών. Ε, Κλείνω το κατάλογο των ομιλητών. Κανείς άλλος? Α, μάλιστα. Ο Κρίς Ντέιβις είναι επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πέθαναν άνθρωποι λόγω της κρίσης αυτής. Και όλοι θα πρέπει να συλλεπιθούμε τις οικογένειες και όλους ε, όσους ε, ακόμα ε, υποφέρουν. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω και τον Επίτροπο όταν παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά πρέπει να αισθάνεστε τελείω αβοήθητο. Το ερώτημα είναι πώ θα εξαγάγουν τα διδάγματα αυτά και ποια διδάγματα θα πρέπει να είναι αυτά. Δεν θα μπορέσουμε, δεν θα είναι παράδεκτο να προσπαθήσουμε να υποσκελίσουμε, να υπονομεύσουμε τις εθνικές αρχές. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα υπάρχει κριτική, αλλά το πιο δύσκολο είναι να πούμε ότι θα έπρεπε να έχει να γίνει. Ωραία λοιπόν, να αναζητήσουμε τα διδάγματα. Το θέμα μπορεί να είναι απλά η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Νόμιζα ότι η ΕΦΣΑ θα έπρεπε να αποτελεί κεντρική αρχή για τέτοια θέματα και τελικά φαίνεται ότι εμπλάκηκε, ε, εμπλάκησε σε μετέπειτα στάδιο. Δεν θα έπρεπε να κάνει κάποιες τέτοιες μελέτες, αναλύσεις. Νομίζω ότι η Εύσα είχε ε, μια τέτοια, ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν άκουσα καθόλου όμως το όνομα της Εύσα καθ' την κρίση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Η Εύσα στην Πάρμα, πόσο γρήγορη ήταν η αντίδρασή της. Ήταν η σωστή υπηρεσία. Η Λίντα Μακέβαν. Ευχαριστώ, Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που συνεχίζονται θα ήθελα να σας ρωτήσω, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην ανείχνευση της πηγής και την αναζήτηση ιατρικών λύσεων. Εκεί θα πρέπει να εστιαστεί η συνεργασία. Αναφέρατε ότι το γιατί θα συζητηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα. Γιατί συνέβη αυτό, από πού προήρθε το μικρόβιο αυτό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Συνδύθηκα με την ε, σχετική αρχή τον είπα και μας είπαν ότι αυτά δεν είναι περίεργα, δεν είναι τα προβλήματα αυτά, δεν είναι ασυνήθιες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, η Ευρώπη δεν είχε ως τώρα προβλήματα με τα λαχανικά και τα φρούτα, με τα προκυπευτικά. Ξέρουμε τι προκαλεί αυτά τα προβλήματα στις ήπα. ξέρουμε τι προκαλεί τέτοια προβλήματα με τέτοια βακτήρια, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ποιος μίλησε με ποιον, το θέμα δεν είναι μόνο η διαδικασία, το θέμα είναι, έχει να κάνει με τη γεωργία. Κάποιοι συνάδελφοι μας είπαν ότι είχαν γίνει πριν από κάποια χρόνια κάποια συζήτηση, συζητήσεις για τη χρήση λιπασμάτων στην γεωργία. Ποια είναι η πηγή κανονικά του E. coli. Σήμερα εξακολουθούν να πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά στο μέλλον μπορεί να υπάρχουν και μαθήματα που πρέπει να εξαγάγουμε για την πολιτική, μακροπρόθεσμα, όχι μόνο ε, μαθήματα για την τεχνική πτυχή της επικοινωνίας, αλλά και για διοργία. Νομίζω ότι για τους πολίτες, αυτό θέλουν να μάθουν οι πολίτες, πώς μπορούν να το αποτρέψουν τον κίνδυνο αυτό, αν πάντα υπάρχει κίνδυνος στα απορροκυπευτικά, τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο αυτό στο μέλλον. Τι γίνεται στις ΗΠΑ, ε, συνεχίζονται αυτά τα περιστατικά, τι γίνεται σε άλλες χώρες, υπάρχουν μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε από άλλες περιοχές. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Μία συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να σας θέσω. Κάτι που με απασχολεί καθόλου τη διάρκεια της, ε, του προστατικού αυτού. Γιατί φαίνεται ότι πήρε τόσο πολύ χρόνο... Α, να περιμένει λίγο να βάλετε και τα ακουστικά σας. Μία συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν να σας κάνω. Φαίνεται ότι πήρε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το πρώτο κρούσμα μέχρι την συγκεκριμένη διάγνωση. Αν δεν έχω άδικο, αν έχω δίκιο στο συγκεκριμένο θέμα, δεν θα έπρεπε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο πόσο γρήγορα μπορούμε να πετύχουμε τη διάγνωση σε παρόμοιο περιστατικό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η πηγή τέτοιων ε, μολύνσεων μετά από δύο-τρεις εβδομάδες. Τα τρόφιμα, από ό,τι ξέρετε, τρώγονται και άρα είναι δύσκολο να εντοπιστούν τέτοιε πηγέ μόλυνσης. Επίσης, αναρωτιέμαι για κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι τα αγκούρια που καλλιεργούνται με σύγχρονους τρόπους μπορεί να ήρθαν σε επαφή με κοπριά. Η βιολογική γεωργία διατρέχει τέτοιους κινδύνους και όχι βιομηχανοποιημένη. Μπορεί να έχει κανείς ε, ε, ό,τι άποψη θέλει για τα είδη της ε, καλλιέργειας, τα είδη γεωργίας, αλλά είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα φυσικό παθογόνο με φυσική αιτία. Άρα, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η διάγνωση. Γιατί διήρκεσε τόσο πολύ, λέει ο Πρόεδρος, μέχρι ότου πατήχουμε τις, ε, διάγνωση. Γιατί στην αρχή πιστεύαμε ότι ήταν τα αγκούρια, μετά πιστεύαμε ότι ήταν τα φύτρα. Αυτό προεκύψε από κάποιους που είχαν πάει σε ένα εστιατόριο και είχαν φάει όλη φύτρα. Ο κύριος Μικολάση. Ε, Ευχαριστώ. λέει ο κύριος Νικολάσικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που σας βλέπουμε εδώ κύριε, ε, κύριε Επίτροπε και που μπορέσατε και αντιδράσατε τόσο γρήγορα. Διότι σε ορισμένους τομείς είναι πολύ δύσκολα να πάρει κανείς γρήγορα αυτές τις αποφάσεις. Θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Εγώ έζησα στον Καναδά μερικά χρόνια και το 2001 προέκυψε μία εμοραγική επιδημία η κόλλη. και τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα ευπαθή διότι χτυπούσε τα, ιδιαίτερα στα νεφρά. Η κατάσταση παρόμοια λοιπόν, αν όχι ίδια. Θα έπρεπε ίσως να ξαναδούμε τις καρτέλες, τις ιατρικές καρτέλες των Καναδών και να δούμε αυτοί τι κάνανε τότε. Είχε βγει τότε στη φορά ένα σκάνδαλο ότι ανθρώπινα περιτώματα τα οχήματα καθάρισης των βόθρων τα έριχναν στο νερό. Δεν θέλω εγώ να πιστεύω ότι έγινε το ίδιο πράγμα στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να κάνουμε έρευνες και προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να εμπλέξουμε τους εμπειρογνώμονες Πολλές φορές αγνοούμε την επιδομιολογία και η ΕΦΣΑ θα πρέπει να έχει πάντοτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί να διαπιστώνει ποια είναι η πηγή της επιδημίας. θα πρέπει τα εργαστήρια να έχουν τις απαραίτητες υποδομές. Διότι όπως έλεγε και ο κύριος ε, Λίζε, στο μέλλον μπορεί να διαπιστώσουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Η επόμενη Μιλιτζιά. Ναι, λέει ο πρόεδρος, περίμενε και την Γερμηνία ε, να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω και τον Επιτροποντάλη που μας έδωσε αυτή την ενημέρωση την... στο Στρασβούργο μέσω των ανακοινώσεων και σήμερα που ήρθε εδώ πέρα να μας παρουσιάσει το θέμα. Δύο θέματα θα ήθελα να τονίσω γιατί πολλά ακούσαμε. Ο Κρίς Ντέιβις και άλλοι αναφέρθηκαν στο ότι θα πρέπει καταρχάς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση σε κατάλληλο επίπεδο, στο εθνικό επίπεδο ή στο κατάλληλο επίπεδο μέσα στην, στο κάθε κράτος. Αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά τέτοια περιστατικά με τρόφιμα, αλλά μπορείτε να μας πείτε αν σας ικανοποίησε ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργήσαν τα δίκτυα ενημέρωσης και πληροφόρησης στην αρχή και ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μήπως ε, ήταν κάτι το οποίο θα θέλετε να έχει συμβεί καλύτερα. Κατά δεύτερον, στην έκθεσή σας που μας αναφέρετε, μιλάτε για τις βελτιώσεις που έγιναν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο στην Ρώμη προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να εντοπιστεί ε, το βακτήριο E. coli στα τρόφιμα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για μία φορά. Θα ισχύσει μακροπρόθεσμα, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη βελτίωση, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως ε, απόρρια του προστατικού αυτού και το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορεί να μας αποτρέψει τέτοιες, ε, από τέτοια προστατικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ε, μια σύντομη παρατήρηση. Την περισμένη εβδομάδα μας είχατε πει ότι θα μιλούσατε με το Συμβούλιο το ίδιο απόγευμα για την επιδημία η κόλλη. Το θέμα είναι ποιος διαχειρίζεται την κρίση, ποιος κυβερνά το πλοίο. Και είπατε ότι θα το συζητούσατε, γιατί πολλέ αρχές ασχολούνται με το θέμα και όταν ε, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει, όπω ξέρουμε. Εσείς προτείνατε κάποια απλοποίηση όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης. Η Γερμανία ασχολείται με το θέμα και από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν πρόθυμη να μοιραστεί τη διαχείριση. Πώς μπορεί να, να διορθωθεί η κατάσταση των κυσμέλων. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, ακούσατε τις ανησυχίες των μελών. με ένα κεντρικό ρόλο για την ΕΦΣΑ, με ένα κεντρικό γραφείο για την καταγραφή και εποπτεία το θέμα της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Τώρα εντάξει δεν είναι αυτή η περίπτωση εδώ, αλλά προκύπτει και αυτό το θέμα. Ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Βασικά, η βασική ανησυχία που άκουσα είναι η ίδια με αυτή που είχα εγώ κατά τη διάρκεια όλες αυτές τις υπόθεσεις της κρίσης. Δηλαδή, ροή πληροφοριών, συντονισμός, που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι εμπειρίες μας στις υπηρεσίες μου δηλαδή κατά τη διάρκεια των ετών αυτών ότι βασικά εδώ θα πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσης ένα κεντρικό σημείο που διαχειρίζεται την κατάσταση και που ενημερώνει για την κατάσταση επίσης. Αν είμαι ευχαριστημένος και ξεκινώ με... γιατί είναι μια από τις ερωτήσεις. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Και τα μηνύματα που έδιναν και που έδινα και στους συναδέλφους στη Γερμανία που πρέπει να πω ότι έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το θέμα, ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο συντονισμό στον τρόπο αντιμετώπισης ε, του προβλήματος. Τώρα, το σύστημα στη Γερμανία είναι όπως είναι. Και εδώ, όσον αφορά τις αρμοδιότητες, Πρέπει να καταλάβουμε την κατάσταση και εδώ να δούμε πώς μπορούμε να αναδιοργανωθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε σε περιπτώσεις όπου θα έχουμε αυτή την πολύ συσχυρές αρμοδιότητες σε επίπεδο κρατηδίων και τοπικών αρχών να υπάρχει τουλάχιστον καλύτερο συντονισμό σε εθνικό επίπεδο που θα τροφοδετεί μετά μια συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς έχει πει και ο Πρόεδρος, η αντίδραση της Ρωσίας και πάλι αποδεικνύει ε, το εξή, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Οποτεδήποτε κι αν συμβεί ένα περιστατικό στα πλαίσια τούτης εδώ της Ευρώπης, της οποίας είμαστε μέρη, ολόκληρη η Ευρώπη θα φέρει το βάρος των συνεπειών των ενεργειών μας. Ακόμα και όταν κανείς ε, είναι λοιπόν πολύ ε, αυστηρό όσον αφορά τι αρμοδιότητέ του, θα πρέπει να καταλάβει ότι οι επιπτώσει είναι για όλου τελικά. Και άρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο συμπαγής ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έστειλα και το οποίο μετέφερα και στην Γερμανία όταν πήγα εκεί για να μιλήσω με τους υπουργούς ε, των, των κατεδίων και τους ομοσπονδιακούς ε, υπουργούς και πήγα να μιλήσω για το τι συνέβαινε σε αυτή τη φάση. Και πάλι επικοινωνία. Αν γίνεται κατάλληλο συντονισμός, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κάποια λάθη που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί ή όπως σας πούμε όταν αναφέραμε το ίδιο το, το όνομα μιας χώρας για την προέλευση των ε, γκουριών κτλ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε αυτό. Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε μία πολιτική τάξη που να είναι αντίθετη στους κινδύνους. Ε, πρέπει να αναλάβουμε ρίσκα κάποιες φορές και να είμαστε διαθέσιμοι γι' αυτό. Ποια είναι λοιπόν τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε ε, και που αποκομίζουμε. Ένα από αυτά είναι το βασικό είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να βελτιώσουμε την πτυχή της επικοινωνίας. Και πάλι εδώ, το θέμα δεν είναι μόνο το πρόβλημα της μακράς αλυσίδας επικοινωνίας, όπως αναφέρατε ορισμένοι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Όχι ο υπουργό του κρατηδίου να πει το τάδε, ο υπουργό ενός άλλου κρατηδίου να πει το δίνα και ο υπουργό υγείας Γερμα... Γερμανίας να πει άλλα και στο Συμβούλιο να υποθούν άλλα. Αυτός ο συντονισμός πρέπει να υπάρχει. Εγώ δεν πιστεύω πως υπήρχε μακριά λυσίδα επικοινωνίας. Όχι, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε έλλειψη συντονισμού. Τώρα, η ΕΦΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας των Τροφίμων, ήταν έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της η ΕΦΣΑ. Πολύ γρήγορα. Τελικά όμως μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο μπόρεσε η ΕΦΣΑ να λειτουργήσει στη Γερμανία. Και αυτό θα πρέπει να πω ότι η συμβολή που έκανε το προσωπικό της ΕΦΣΑ για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών διαδικασιών ήταν εξαιρετικά χρήσιμες και ωφέλη μας. Η ΕΦΣΑ λοιπόν ενέργησε τάχιστα, ήταν έτοιμη να κινηθεί πολύ γρήγορα, αλλά και πάλι είναι θέμα αρμοδιοτήτων εκεί, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα άλλο και αυτό θα πρέπει να είναι άλλο ένα μάθημα, που άλλο ένα δίδαγμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε στο μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε μια πλήρη ανάλυση των όσων ε, του τι μάλλον οδήγησε αυτό το παθογόνο στην τροφική αλυσίδα. Καταρχήν, και από ό,τι ακούω και πάλι, είναι θέμα ενός ε, δηλαδή, είναι θέμα μόλυσης από περιτώματα. Τώρα, αν ήταν σε συγκεκριμένο αγρόκτημα που εντοπίσαμε, αν ήταν στο πλοίο που μετέφερε τους σπόρους στο συγκεκριμένο αγρόκτημα, Όλα αυτά θα πρέπει να τα ανεχνεύσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένα τομέα που θα εστιάσουμε την προσοχή μας, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό να βρούμε την αρχική πηγή. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί προχωρήσαμε τόσο πολύ στο να εξασφαλίσουμε την πηγή ε, της, που προκάλεσε την μόλυνση. Γιατί κάποιες φορές ούτε αυτό δεν είναι δυνατόν. Ούτε, αλλά και πάλι δεν πρόκειται να επαναφερθούμε στις δάφνες μας, θα κινηθούμε πολύ πολύ πιο πέρα για να προσπαθήσουμε να βρούμε την πραγματική αιτία. Επίσης θα κάνουμε μελέτη για το συγκεκριμένο παθογόνο ή μάλλον ε, ομάδα παθογόνων ε, τις εμπειρίες από τη Καναδά, τη ΣΥΠΑ θα τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε πιο λεπτομερή επιστημονική ανάλυση αφού του είδους του προβλήματος για το εργαστήριο της Ρώμης είναι ένα από τα εργαστήρια κατεξοχήν εργαστήρια με τα οποία συνεργαζόμαστε ε, και χρηματοδοτούμε για συγκεκριμένα θέματα και εδώ βρισκόμουν στη Ρώμη ούτως ή άλλως και θεώρησα ότι έπρεπε να επισκεφτώ αυτούς τους ανθρώπους που μας κάνουν περήφανος νομίζω γιατί μπόρεσαν τόσο γρήγορα να ε, εντοπίσουν το πρόβλημα και να καταλάβουμε ακριβώς και πώς ε, λειτουργεί το πράγμα. Αυτή είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση λοιπόν, είναι μια, ένα ερευνητικό εργαστήριο το οποίο ασχολείται με την έρευνα σε τέτοια θέματα. Δεν φτάσαν σε αυτό το αποτελέσμα σαν μια νυχτή, ήταν αποτέλεσμα ε, διαδικασιών που είχαν ξεκινήσει από παλιότερα για το πώς μπορούν να επιτευχθούν τέτοια πράγματα. Τελικά δηλαδή είδαμε ότι μπορούσαν να ε, εστιάσουν στο συγκεκριμένο θέμα και θα εκδοθεί και συγκεκριμένη έκδοση στις 18 ε, Νοεμβρίου που είναι η ημέρα κατά των βακτηριδίων. Σας ευχαριστώ Επιτρόπε. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση. Επικεντρωθήκαμε σε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία και λαμβάνουμε γνώση των δραστηριοτήτων σας και των ενεργειών των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών. Η Επιτροπή μας θα παρακολουθήσει λοιπόν τη συζήτηση και τα περιστατικά και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι η τελευταία νόσος που γνωρίζει η Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να διδαχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και να βελτιώσουμε τη στάση μας για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε και πάλι που παρευρεθήκατε εδώ. Αύριο το πρωί στις 9 ξεκινάμε με την συνεδρίαση των συντονιστών.